Καλημέρα σας. Συγγνώμη, η ελληνική καμπίνα. Είχαμε τεχνικό πρόβλημα και πρέπει να αλλάξουμε καμπίνα. Έχουμε λοιπόν αυξημένη υποστήριξη από τον προπολογισμό και αντίστοιχα αιτήματα. Σε ό,τι αφορά τώρα τη λεγόμενη δήλωση αξιοπιστίας για την αξιοπιστία των λογαριασμών. Σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης χρειάζεται προσοχή γιατί η λογιστική μέθοδος που χρησιμοποιούμε στους λογαριασμούς μας στην Ευρώπη δεν ισχύει για όλες τις συμβάσεις. Το γνωρίζει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει την πρόθεση από το 2009 και μετά, το οικονομικό έτος 2009, να αλλάξει, να θεωρήσει τον τρόπο με τον οποίο γίνονται. Σε ό,τι αφορά τώρα την αξιοπιστία των υποκειμένων συναλλαγών, δυστυχώς οφείλω να τονίσω ότι παρά την επέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να διευκολυνθεί η διαδικασία αυτή, το ελεκτικό συνέδριο δεν πήρε όλες τις απαραίτητες ε, πληροφορίες σε ό,τι αφορά 10 συναλλαγές από διεθνείς οργανισμούς, Αφρικανική Ένωση, Παγκόσμια Τράπεζα, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Για το λόγο αυτό το ελεκτικό συνέδριο δεν ήταν σε θέση να ελέγξει λογιστικά πλήρως αυτές τις οικονομικές ε, συναλλαγές και δεν έχει ε, την ευκαιρία να εκφράσει άποψη για 119 εκατομμύρια που είναι 6,7% του ετησίου προϋπολογισμού των ετησίων δαπανών καλύτερα για το ETF. με αυτή την εξαίρεση γενικά θεωρούμε ότι είναι κανονικές και νόμιμες οι δαπάνες. Οι υποκείμενες όμως συναλλαγές σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ελέγχθησαν. Τώρα, πρέπει να πούμε ότι σε πολλές περιπτώσεις έχουμε μη ποσοτικά μετρήσιμα σφάλματα στη μακροοικονομική βοήθεια. Τρεις τέτοιες περιπτώσεις εντόπισε το ενακτικό συνέδριο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εξήγησε σωστά ε, αν ήταν ε, ε, σωστή, διαφανής και χρηστή η διαχείριση στη δημόσια διοίκηση κάποιων κρατών. Ωστόσο, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, το ελεκτικό συνέδριο βρήκε ότι Βελτιώνεται η συμμόρφωση προς τα κριτήρια Κοτονού για τους στόχους κυρίως της ε, χιλιετίας και της αντίστοιχης συμβάσης. Αυτό έχει να κάνει και με το δέκατο ε, Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης που έχει μια νέα συμφωνία χρηματοδότησης και διαπιστώνει και το ελεγκτικό συνέδριο ότι ε, επιτελείται πρόοδος εκεί. Θα ήθελα μόνο να σας πω ότι έχουν γίνει επιτυχείς διαπραγματεύσεις και συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να είναι πιο διαφανής η διαδικασία μακροοικονομικής βοήθειας. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν συμφώνησε να ε, βάλει κάποιους ε, ελάχιστου όρους. Συμφωνεί ότι χρειάζονται βελτιώσεις, όπως λέγει και το ελεκτικό συνέδριο, για την υποστήριξη των αποφάσεων που έχουν ήδη ληφθεί. Σε ό,τι αφορά τις πληρωμές, ε, φρονεί το συνέδριο ότι έχουμε 2 ε, με 5% ε, υλικά σφάλματα. Αντίστοιχα με τα προηγούμενα έτη, επισχύουν για την επιλεξιμότητα. Έχουμε, ας πούμε, δαπάνες που έχουν καταβληθεί εκτός της προβλεπόμενης περίοδου, λεξιπρόθεσμα ή με αντικείμενα που δεν είναι επιλέξιμα. Ας πούμε δεν είχαμε τιμολόγια. Και άλλες σημαντικά συναντευτικά παραστατικά. Και φυσικά προβλήματα στους υπολογισμούς, σφάλματα σε υπολογισμούς και ε, όπως σας είπα μη ποσοτικά μετρήσιμα ε, ε, ορατότητα, διαφάνεια, δημόσιες συμβάσεις, τραπεζικές εγγύησεις ε, σε ό,τι αφορά τη μακροοικονομική βοήθεια, ε, πολλές φορές δεν εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις οι όροι που συνδέονται με την καταβολή των πληρωμών, στοιχεία που δεν συλλέγονται, στοιχεία ε, απαρχιωμένα που δεν μπορούν να επιτρέψουν την καλή χρηστή διαχείριση και την περίοδο αναφοράς για να μετρούμε το, πόσο λειτουργούν οι δείκτες. Αυτά είναι σφάλματα και δείχνουν αδυναμίες σε διάφορα επίπεδα στα συστήματα ελέγχου και εποπτείας. Και επιτρέψτε μας να σας αναφέρω τα πιο σημαντικά. Πρώτον, ο εσωτερικό λογιστικό έλεγχο συχνά είναι ασθενή. Ε, μιλώ για τους οργανισμούς που επιφορτίζονται με την ε, εκτέλεση αυτού του έργου. Ε, ε τα συστήματα χρηματοδότησης και τήρηση λογιστικών βιβλίων δεν εξασφαλίζουν ότι η δαπάνη καταγράφεται και κοινοποιείται σωστά. Σε άλλες περιπτώσεις η ποιότητα του ελέγχου που γίνεται από κάποια εποπτική αρχή επίσης χωλαίνει σε μεμονωμένες συμβάσεις έργου. Και ένα τελευταίο που είναι όμως σημαντικό, ε, συχνά υπάρχει πρόβλημα κυριότητας ιδιοκτησίας ε, στις περισσότερες υπηρεσίες διατακτών ε, στα κράτη αυτά. Οπότε είναι και η έλεγχη ε, ελλειπής. Γενικά, επειδή υπάρχουν αυτές οι αδυναμίες και τα προβλήματα, ε, έχουν λάβει μέτρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να τα αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα με υποχρεωτικούς λογιστικούς ελέγχους και επαληθεύσεις ε, των δαπανών πριν κλείνουν τα έργα και ολοκληρώνονται. Επίσης υπάρχει η τεχνική βοήθεια στις συμβάσεις ε, για να μπορούν καλύτερα να ελέγχουν οι αρμόδιες αρχές. Το 2008 η Europe Aid ε, ζήτησε ε, καλύτερες κατευθυντήριες γραμμές και μέσα επικοινωνίας για να αντιμετωπιστούν παγκοσμίω αυτές οι αδυναμίες και να ε, ωφεληθούν τελικά οι τελικοί δικαιούχοι και οι εκτελεστικοί οργανισμοί. Κυρίες και κύριοι, το 2008 η EuropeAid συνέχισε να βελτιώνεται σημαντικά ως προς το σύστημα ελέγχου και εποπτείας της. Άρχισε να χρησιμοποιεί τους νέους όρους αναφοράς για το λογιστικό έλεγχο και ένα διαχειριστικό νέο σύστημα που κανονικά θα πρέπει να βελτιώσει τη δυνατότητα να ελέγχει, να σχεδιάζει, να αναλύει και να παρακολουθεί τις ε, συστάσεις και τα ευρήματα. Η αιτήσια έκθεση δραστηριοτήτων της EuroPaid είναι καλύτερη, είναι πιο κατατοπιστική και πιο σαφής και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι χρησιμοποιούνται καλύτερα οι ποσοτικοί δείκτες. Η Europe Aid έχει κάνει μια ευρεία στρατηγική ελέγχου για να έχουμε πιο ε, αποτελεσματικούς ελέγχους, όπως σας είπα. Για να ε, συμβάλλει προς τη κατεύθυνση αυτή, το ελεκτικό συνέδριο κάνει πολλές συστάσεις, εξίσου σημαντικές όλες. Επιτρέψτε μου όμως να σας αναφέρω τις εξής. Πρώτον, ε, εκ των προτέρων έλεγχοι που θα πρέπει να βελτιώνονται, εστιάζοντας σε βασικούς κινδύνους. Δεύτερον, ετήσιες εκθέσεις ε, λογιστικού ελέγχου θα πρέπει να προετοιμάζονται με τρόπο πιο ρεαλιστικό και ε, αναλύοντας το πραγματικό κίνδυνο. Τα ετήσια αυτά προγράμματα θα πρέπει να εφαρμόζονται με τρόπο καλό και να παρακολουθούνται έτσι ώστε εγκαίρως να εντοπίζονται αποκλήσεις και να ανοιχνεύονται ε, τα προβλήματα για να διορθώνονται. Χρειάζεται πιο αναλυτική λοιπόν παρακολούθηση και συνέχεια ε, των αποτελεσμάτων αυτών. Η Europaid θα πρέπει να αναθεωρεί ε, το σύστημα ελέγχου εκ των υστέρων έτσι ώστε να επεκταθεί ε, το πεδίο εφαρμογής των ελέγχων αυτών. Και τέταρτο, σε ό,τι αφορά τη χρηματοοικονομική βοήθεια, τη μακροοικονομική βοήθεια, η Europaid θα πρέπει να συνεχίσει ε, τις προσπάθειές της για την ε, επιλεξιμότητα με τρόπο διαρθρωμένο και σωστό. Ε, να έχει ένα καλό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων η δικαιούχος χώρα με προβλέψιμα χρονοδιαγράμματα και με δέσμευση των χωρών που συμμετέχουν για την εφαρμογή του προγράμματος αυτού. Θα πρέπει επίσης όλες οι μελλοντικές συμφωνίες χρηματοδότησης να έχουν μια ευρεία και σαφή βάση για τη συμμόρφωση με τις συνθήκες και τις όρους πληρωμής. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω ολοκληρώνοντα τι υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εξαιρετική συνεργασία και υποστήριξη και τι πολύ καρποφόρε συζητήσει που είχαμε όταν κάνουμε παρατηρήσεις. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω για ε, την επικοδομητική ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις συστάσεις του Ελεκτικού Συνεδρίου. Ε, έχουν ήδη ασχοληθεί και αντιμετωπίσει με όλα τα προβλήματα που εντοπίσαμε στην έκθεσή μας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Είναι παρόν και ο Επίτροπος ε, Κάρλ Ντεγκούτ, υπεύθυνο για την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια, στον οποίο δίνω και το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριοι συγητές, ε, μέλη της Επιτροπής, ε, μέλη του Ελεκτικού Συνεδρίου, κυρίες και κύριοι, όπως γνωρίζετε, ανέλαβα καθήκοντα ε, Επιτρόπου υπεύθυνη για την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια στα μέσα Ιουλίου. Παρά το γεγονός ότι εργάζομαι πάνω σε αυτό το θέμα ε, ελάχιστο χρονικό διάστημα, εστίασα την προσοχή μου στην ε, βελτίωση της ποιότητας της ανθρωπιστικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι εδώ σήμερα συζητούμε πώς μπορούμε να κάνουμε την ανθρωπιστική βοήθεια πιο αποτελεσματική, πιο διάφωνη και πιο εύκολη στη διαχείρισή της. Έχουν καταγραφεί πολλά στοιχεία ε, που αφορούν στη διαχείριση του ε, Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης. Έχουμε διαπιστώσει αρκετές ελλείψεις και θεωρούμε ότι υπάρχει και περιθώριο βελτίωσης. Ε, στο λίγο διάστημα που εργάζομαι στο θέμα αυτό, πρέπει να πω ότι έχω εντυπωσιαστεί από τη δουλειά που κάνουν οι υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρά το γεγονό ότι, όπω είπα και πριν, έχουμε περιθώριο βελτίωση. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειε και δεν θα σταθώ σε όλα ένα προ ένα τα σημεία τη έκθεση. Θα ήθελα να σταθώ σε κάποια πιο πολιτικά σημεία, τα οποία θεωρώ ότι χρήζουν λίγο περισσότερη προσοχή. Όσον αφορά στην ανθρωπιστική βοήθεια και στην αποτελεσματικότητά τη, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει περίπου το 60% τη επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια ε, παγκοσμίω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν ο τρίτο μεγαλύτερο δωρητή το 2008. Οι νέε δεσμεύσει από πλευρά κρατών μελών και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν αυξηθεί από τι 30.000 το 2003 στι 40 με 50.000 το 2005 και είναι πάρα πολλές για να είναι αποτελεσματικές. Έφυξα το θέμα αυτό στο Συμβούλιο τον περασμένο μήνα. Έγιναν κάποιες καλές προτάσεις, αλλά αν θέλουμε να βελτιώσουμε τον ογετικό ρόλο που έχουμε στην αναπτυξιακή βοήθεια, θα πρέπει να αποδώσουν και καρπούς όλες οι δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει. Η σχέση μεταξύ δωρητών και ε, η προσπάθεια για καλύτερη κατανομή των πόρων είναι απλά παραδείγματα που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Επίσης πρέπει να μειωθεί το διαχειριστικό και το γραφειοκρατικό κόστος και επίσης θα πρέπει να ε, ξέρουμε ποιος είναι υπόλογος γιατί σε εσωτερικό επίπεδο. Στη διάρκεια του 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ε, νέες ε, ε, δραστηριότητες υποστήριξης βάσει του 10ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης σε περισσότερες χώρες ε, με βάση τους στόχους της χιλιετίας. Είχαμε μακροπρόθεσμους ε, όρους, περισσότερη υποστήριξη σε χώρες οι οποίες έχουν καλό μητρό. Για να είναι όμως τα πράγματα πιο ασφαλή θα πρέπει να υποστηρίξουμε και το ρόλο των τοπικών κοινοβουλίων, της κοινωνίας των πολιτών, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, υποστήριξη προς όλα τα θεσμικά όργανα, στις οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στα θέματα αυτά και ε, να δούμε τι γίνεται και με τις δαπάνες. Χαιρετίζουμε και τις παρατηρήσεις του Συμβουλίου για την υποστήριξη από πλευράς προϋπολογισμού. Η έκθεση που έχουμε ε, αναφέρει τα πρόοδο που έχει γίνει το 2008 έχει δοθεί καλύτερη διάρθρωση στην πρόσφατη υποστήριξη του προπολογισμού και επίση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει υπόψη την και τι συστάσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίε προέκυψαν από την απαλλαγή του 2007 για την ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια για τη διαχείριση και, ε, και τι εκθέσει για τον προπολογισμό. Αν θέλουμε να έχουμε την αναπτυξιακή βοήθεια ε, με πιο αποτελεσματικό τρόπο θα πρέπει να μειωθεί και το γραφειοκρατικό και διοικητικό κόστος. Δαπανώνται τεράστια ποσά ετησίως για να βελτιωθεί η ανθρωπιστική βοήθεια και η αναπτυξιακή βοήθεια και οι εξωτερικές δράσεις εφαρμόζονται σε ένα περιβάλλον υψηλού κινδύνου οι χώρες εταίροι πολύ συχνά έχουν υποανάπτυκτα διοικητικά και γραφειοκρατικά συστήματα και φυσικά ε, υπάρχουν ε, καθημερινές διαμάχες στο καθημερινό μας περιβάλλον εργασίας. Πρέπει να λάβουμε μέτρα εποπτείας για να μπορέσουμε να μετριάσουμε τα αποτελέσματα αυτά και να υπάρχει και αλλά το γεγονός ε, ότι μπορεί να υπάρχει πάντα ένα περιθώριο σφάλματος πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. ένας έλεγχος που έγινε το 2008 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη κάλυψε και την Αγκόλα η οποία βρισκόταν σε ε, φίλια διένεξη και καταλαβαίνετε ότι ήταν πολύ πιο δύσκολη η έλεγχη. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να ζητήσω από αυτόν που θα με διαδεχθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά να ζητήσω και από εσά ε, να λάβετε υπόψη σας πολύ ε, σοβαρά το θέμα των κινδύνων που προκύπτουν από τα σφάλματα θα πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική ε, για την αναπτυξιακή βοήθεια, την οποία σκοπεύει να ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή του χρόνου και θα πρέπει να μας βοηθήσει στο έργο μας. Θα πρέπει να γίνουν σημαντικές βελτιώσεις σε αρκετούς τομείς, όπως έχει αναγνωρίσει και το ελεγκτικό συνέδριο και όλα αυτά μπορεί να μην είναι τόσο προφανή ε, από την πρώτη στιγμή. Καταλαβαίνω ότι το ελεγκτικό συνέδριο ε, προσπαθεί να μας ενθαρρύνει να κάνουμε περισσότερα. Ο εξορθολογισμό όμως τη προσέγγιση που έχουμε για τους ελέγχου είναι πολύ ενθαρρυντικός και θα, ε, θέλαμε να συνεχίσουμε, πιστεύουμε ότι θα έχουμε πολύ καλύτερες βελτιώσεις. Θα ήθελα εντάχει να σταθώ και λίγο στο υπόλοιπο τμήμα του χαρτοφυλακίου μας, την ανθρωπιστική βοήθεια. Η ΕΚΟ έχει κάνει πολύ σημαντικές βελτιώσεις το 2008 για να αυξήσει την κάλυψη που έχει στους ελέγχους και αυτό ως απάντηση στις προηγούμενες επικρίσεις ε, και χαίρομαι που διαπιστώνω ότι και σε αυτή την περίπτωση αναγνωρίζεται η προσπάθειά μας από το ελεγκτικό συνέδριο. Κύριε Πρόεδρε, μέλη της ε, Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού, ε, μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σε ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Το λόγο στον πρώτο εισηγητή μας, τον κύριο Λιμπεράσχη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο ε, Ουσκεβιτς του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τον Επίτροπο Κάρολ Τιγκούχτ για τη συζήτηση και την παρουσίαση του θέματος για το σημαντικό αυτό θέμα. Στην αρχή σχόλια και μετά ερωτήσεις. Ανάλυση κινδύνου. Οι πιο φτυχές χώρες έχουν πιο επίγουσα ανάγκη. Είναι δυνατόν να αποφευθεί ο κίνδυνος, αλλά να μειωθεί ο κίνδυνος είναι δύσκολο έργο. Ξέρω ότι η Κομισιόν θα έπρεπε να αναλάβει σημαντική προσπάθεια για να πετύχει συμφωνία στα Ηνωμένα Έθνη, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και μερικέ μη κυβερνητικέ οργανώσει να συνεργάζονται. Κύριε Πίτροπε, κατά τη γνώμη μου, ο ρόλο σα είναι να αποφύγετε τα διάφορα παράπονα που ακούσαμε από τον κύριο σκέψη για το 9,3% των χρημάτων που δεν καλύπτονται από τους ελέγχους. Βέβαια υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες πράξεις, πάρα πολλές χώρες. Έχει σημειωθεί η πρόοδος. Αν το, μεσ, ε, το μήνυμα είναι να γίνει πιο ορατή η Ένωση και πιο ορατή ως μια πολιτικά φιλική χώρα για τις φτωχές αυτές περιοχές του κόσμου και δύο ερωτήσεις. Η κυρία Ενέσα Γιάλα Σέντερ θα κάνει πολύ περισσότερες ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση. Η βελτίωση στις εξωτερικές δαπάνες είναι θετική. Βελτίωση 40%. Πώς το εξηγεί όμως η Κομισιόν αυτό και τι περαιτέρω περιθώριο βελτίωσης υπάρχει. το 2009 να περιμένουμε βελτίωση μέχρι 40%. Δεύτερη ερώτηση. Τι πρόοδος σημειώθηκε σε κοινή εποπτεία των δαπανών για τις εξωτερικές δράσεις. Τα Ηνωμένα Έθνη και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Τι να περιμένουμε ως βελτιώσεις. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Και η κυρία Αγιάλα Σέλτερ, δεύτερη συγκήτρια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω για όλα όσα ακούσαμε πριν από λίγο. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν και τον εκπρόσωπο του ελεγκτικού συνεδρίου Νομίζω ότι είναι πολύ καλή συνεργασία και ήταν πολύ χρήσιμες οι επισημάνσεις του και ο διάλογος ε, μέσω του οποίου μου έδωσε και όλη τη βιβλιογραφία ε, και προσπάθησα λίγο να οργανωθώ χάρη και στην βοήθεια της γραμματείας της Επιτροπής μας ε, με διευκόλυνε σε πάρα πολύ δύσκολα πράγματα Υπάρχει ένας τεράστιος ωκεανός ε, δεδομένων και στοιχείων και ε, νομίζω ότι η βοήθεια του ελεγκτικού συνεδρίου ήταν ο φάρος που φώτισε ε, τη δουλειά μου και ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι βρισκόμαστε ενώπιον μιας κατάστασης ε, όπου ακούμε τον κύριο Ντεγκούχ, το οποίο έκανε μια πάρα πολύ καλή δουλειά σε τέσσερις μήνες ε, που έχει αναλάβει το χαρτοφυλάκιο αυτό αυτή τη στιγμή είναι υποχρεωμένος να δώσει ε, λόγο σε εμά στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού για όλη τη διαχείριση που έκανε ο κύριος Λουί και ε, ούτως ή άλλως είναι πρώτον πυλών για αλλαγή χαρτοφυλακίου θα αναλάβει τα θέματα εμπορίου όπως ξέρετε και ελπίζω Όλο ο κόπο και όλη η ευαισθητοποίησή του τους τελευταίους τέσσερι μήνε, μήνες, ε, ούτως ή άλλως ήταν ε, υπουργό ε, στο Βέλγιο πριν από αυτό, αλλά το θέμα της ανθρωπιστικής βοήθειας και ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα σας βοηθήσει πολύ στο νέο σας χαρτοφυλακείο που είναι θέματα εμπορίου που αν θέλετε είναι η άλλη όψη του νομίσματος για τις εξωτερικές σχέσεις με τον υπόλοιπο κόσμο, τόσο εντός όσο και εκτός ε, συνόρων. Σας εύχομαι λοιπόν ότι καλύτερο στη νέα σας ε, καριέρα, αλλά επειδή αυτή τη στιγμή είστε ακόμα υπεύθυνο σε θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας και ανάπτυξης, ε, που όπως ε, και εσείς είπατε είναι ένα από τα πιο αγαπητά θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι είναι παγκόσμιος εταίρος ε, και θέλει να είναι παγκόσμιος εταίρος γι' αυτό λοιπόν θα έλεγα ότι είναι και ένα από τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας που προσδίδουν περισσότερη καινοτομία όχι μόνο γιατί είμαστε ο πρώτος δωρητής παγκοσμίως αλλά και γιατί Υπάρχει ανάπτυξη, φαντασία, δημιουργικότητα από πλευρά υπηρεσιών. Εγώ τα παρακολουθώ πάντα αυτά τα θέματα και ε, πάντα ε, μπορούμε να προσφέρουμε κάτι για την επίλυση συγκρούσεων, για ε, να προσπαθήσουμε να έχουμε κάποια στοιχεία ε, για κάθε κράτος μέλος και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε εκεί όπου υπάρχουν προβλήματα. Πρόκειται λοιπόν για κάτι το οποίο είναι πολύτιμο και το οποίο όπως είπε και ο συνάδελφος Λιμπεράσκη θα πρέπει να το βελτιώσουμε διότι οι πολίτες στα λίγα θετικά πράγματα που αναγνωρίζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμπεριλαμβάνουν και την αναπτυξιακή βοήθεια και τη δυνατότητα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, συνδράμει άλλες χώρες, κυρίως χώρες που έχουν τις περισσότερες δυσκολίες. Να ευχαριστήσω λοιπόν και για όλη την ε, προσπάθεια που έγινε για αυτό το διάλογο. Ε, υπήρχαν κάποιες φυσικά διαφορές απόψεων ε, μεταξύ Ελεγκτικού Συνεδρίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς τα θέματα τα οποία χρήζουν βελτίωση. Εγώ χαίρομαι που το Ελεγκτικό Συνέδριο που μας λέει ότι θεωρεί ότι είναι επιτυχία αυτή η πορεία ε, μέχρι την έκθεση και επίσης στις ε, απαντήσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπήρχαν ήδη προτάσεις για τροπολογία να έχουμε πιο επίσημα μέσα τα οποία θα είναι πιο καλά για τους ελέγχους, ε, κυρίως για τους εκτοπροτέρων ελέγχους που νομίζω ότι είναι η έλεγχοι που είναι οι πιο αποτελεσματικοί. Διαπιστώνω ότι το ελεγκτικό συνέδριο πλέον επικεντρώνεται περισσότερο στους εκ των προτέρων ελέγχους και χαίρομαι, θα ήθελα να μας πει όμως λίγο περισσότερα πράγματα το ελεγκτικό συνέδριο. Ο διάλογος αυτός είναι μία από τις πτυχές που θέλει να ε, προωθήσει περαιτέρω η Επιτροπή μας ε, και με τα δύο θεσμικά όργανα, διότι είναι από τα πράγματα που μας έχουν ζητήσει και οι πολίτες. Να πω επίσης ότι βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή, διότι μόλις έχει ξεκινήσει η εφαρμογή της νέας συνθήκης, Υπάρχει τη εκπρόσωπος για τα εξωτερικά ε, θέματα και χαιρετίζουμε και τον διορισμό της, αλλά υπάρχουν και μια σειρά από πτυχές οι οποίες ε, δημιουργούν ε, μεγάλα ερωτηματικά πώς θα διαρθρωθεί η διαδικασία λήψης απόφασης και όλη αυτή η δομή και η διασύνδεση μεταξύ Γενικής Διεύθυνσης Ρελέξ και Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και το νέο θέμα της ευρωπαϊκής διπλωματίας το οποίο θα ξεκινήσει ε, πλέον και θα διαδραματίσει εξίσου σημαντικό ρόλο. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα ε, ο Επίτροπος επειδή αυτή τη στιγμή έχει αυτή την ελευθερία αν θέλετε, έχει ένα ε, σύντομο διάστημα αρκετά έντονο διαχείρισης και θα αναλάβει τώρα ένα νέο χαρτοφυλάκιο ε, ίσως θα μπορούσε να μας πει ε, με την πείρα που έχουμε τώρα ποια είναι αυτά τα πιο σημαντικά σημεία αυτής της έκθεσης η οποία πάντα δημιουργούσε ε, διενέξεις για το ποιος ε, παίρνει τι, ποιος συντονίζει τι, τι γίνεται με προσωπικό, τι γίνεται με τους στόχους ε, μεταξύ Γενικής Διεύθυνσης Ρελέξ και Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης. Ε, κυρίως σε σχέση και με αυτό το νέο ορίζοντα που έχουμε μπροστά μας πλέον. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω αν μπορεί ο κύριος Δεχούκ να μας πει κάποια πράγματα παραπάνω. και επίσης να σταθώ λίγο και στα πιο συγκεκριμένα σημεία που αφορούν τη δική μας την ε, διαδικασία, την απαλλαγή για το 2008. Άκουσα και διαπίστωσα και επιτόπου ε, και με τον ε, ε υπεύθυνο του Ελεκτικού συνεδρίου στην αντιπροσωπεία που είχαμε στο Κωσυφοπέδιο όταν ήμουν υπεύθυνη για την έκθεση για τους οργανισμούς τι μπορούμε να κάνουμε με τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση όταν έρχεται σε επαφή με τον προπολογισμό άλλων διεθνών οργανισμών. Ο κύριο ε, Λιμπεράτσκι το είπε σαφώ και θα είναι μία από τι ερωτήσει που υποστηρίζω και εγώ. Θα ήθελα να ξέρω τι γίνεται με αυτέ τι δυσκολίε. Είναι σκοτεινό το τοπίο και το ελεγκτικό συνέδριο δεν καταφέρνει να πάρει την απαραίτητη τεκμηρίωση. Και αυτό είναι σκανδαλώδε. Επίση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό τον κοινό προγραμματισμό ε, δεν ξέρω κατά πόσον μπορεί να υποχρεώσει τους οργανισμούς όχι να ενοποιήσουν, αλλά τουλάχιστον να οργανώσουν τον τρόπο συνεργασίας, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δικαίωμα να ξέρει τι γίνεται με τα σχεδόν 200 εκατομμύρια βοήθειας ε, που δίνει σε συνεργασία με αυτούς τους διεθνείς οργανισμούς. Και επίσης θα ήθελα με βάση αυτά που θα κάνουμε για την απαλλαγή αυτή να δημιουργηθούν και κάποιοι τρόποι ε, να είμαστε λίγο πιο παραγωγικοί. Εξακολουθεί να είναι μελανό αυτό το σημείο και όπως είπε και ο κύριος Λιμπεράτσκι, αφορά πολύ σημαντικούς ε, διεθνείς οργανισμούς, τα Ηνωμένα Έθνη, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ε, μιλάμε για οργανισμούς που μπορεί να είναι πιο μακριά μας, αλλά να είναι και μέσα στην καθημερινότητά μας. Και φυσικά επηρεάζει και πολλά πράγματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μαζί με τους συναδέλφους λοιπόν θα πρέπει ίσως να εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο αυτό το πρόβλημα το οποίο γίνεται όλο και πιο σημαντικό. Δεν θέλω καν να φανταστώ τι μας περιμένει πλέον με τα νέα μέσα που θα έχουμε μετά από τη συνεργασία, διότι θα έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική χρηματοδότηση, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υπησέλθει και σε αυτή τη ε, διαδικασία και θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να ελέγξουμε και εκ των προτέρων και εκ των υστέρων και να υποσημοποιηθεί αυτός ο έλεγχος και η συνεργασία ε, των διεθνών οργανώσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μην βρεθούμε και αντιμέτωποι. Μέχρι τώρα τα πράγματα αυτά δεν τα μετρούσαμε, αλλά νομίζω ότι πλέον μπαίνουμε σε πολύ πιο βαθιά ύδατα. Όσον αφορά τώρα στην ε, βοήθεια στον προπολογισμό, πρόκειται για έναν από τους πυλώνες καινοτομίας για την αναπτυξιακή πολιτική Υπήρχαν και εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι, το είπαν και τα δύο όργανα εδώ, και το Ελεκτικό Συνέδριο και το αναγνώρισε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βέβαια έχουμε κάποιες βελτιώσεις, αλλά δεν πάει να είναι αλήθεια ότι υπάρχουν ε, ε, προβλήματα ακόμα και είναι επίσης αλήθεια ότι οι πολίτες τα γνωρίζουν αυτά τα θέματα διότι προβάλλονται στον τύπο τα στοιχεία για το τι γίνεται με την αναπτυξιακή βοήθεια. Κάποιες χώρες ε, έχουν ε, ε, φίλοι σειράξει ή αντιδημοκρατικές διαδικασίες, ο, ο του τους ε, πάσχει με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Πώς μπορούμε λοιπόν να ελέγξουμε από την αρχή μέχρι το τέλος αυτή τη βοήθεια που, που δίνεται ότι οι χώρες οι οποίες λαμβάνουν την αναπτυξιακή βοήθεια Εξακείμενο όχι μόνο του ελέγχου του προπολογισμού, αλλά ε, βλέπουν τι γίνεται και σε πολιτικό και σε κοινωνικό επίπεδο. Νομίζω ότι και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό και θα ήθελα να ρωτήσω κάποια πράγματα από το ελεγκτικό συνέδριο, διότι υπάρχουν μέσα, μπορεί κάποια μέσα να μην είναι τόσο επίσημα, αλλά μπορεί να έχει τη δυνατότητα να κάνει κάποια ακρόαση σε, ένα, ε, σε μια χώρα στην οποία δεν υπάρχει σύγκρουση. Μιλήσαμε και για το επίπεδο αποδεκτού κινδύνου που νομίζω ότι είναι ένα από τα πράγματα τα οποία Με συγχωρείτε, συγκινήθηκα, λέει η κυρία Γιάλα. Σα ζητώ συγγνώμη, λέει ο πρόεδρο. Είμαι δημοκρατικό πρόεδρο, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν πάρα πολλέ παρεμβάσει και επειδή πρέπει να θέσουμε ερωτήσει προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σα παρακαλώ να επιταχύνετε λίγο, γιατί αλλιώ δεν θα έχουν χρόνο οι άλλοι συνάδελφοι να μιλήσουν. Ε, ναι, κύριε πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη. Ε, είχα πάρα πολλέ πληροφορίε, δεν μπόρεσα να είμαι πιο συνοπτική. Να ξαναπώ λοιπόν για άλλη μια φορά αυτέ τι δύο ερωτήσει. Ε, τι γίνεται με τι σχέσει με του διεθνεί οργανισμού και την βοήθεια στον προπολογισμό. Θα μπορούσαν και οι δύο, ε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο, να μα πούνε λίγο πιο συγκεκριμένα πράγματα και τι γίνεται με ένα κάποιο πιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη που μακρηγόρησε. Ευχαριστώ. Δίνω τον λόγο στον Επίτροπο Ντεγκούκ για να απαντήσει στα ερωτήματα των εισηγητών. Thank you, uh, Mr. Chair. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. This, uh, about, uh, how to work, Αυτό το θέμα της συνεργασίας με τους διεθνείς οργανισμούς ε, κάθε χρόνο επανέρχεται βλέπω από τους φακέλους. Και δεν ήταν εύκολο να βρεθεί λύση. Αλλά νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όντως βρήκε μια λύση και συνεχώς προσπαθεί να κινητοποιήσει τους διεθνείς οργανισμούς και τους ε, οργανισμούς του ΟΗΕ και να τους παροτρύνει να έχουν μεγαλύτερη διαφάνεια. Και μία από τις παρατηρήσεις που ακούμε από τους οργανισμούς αυτούς είναι ότι ο βαθμός διαφάνειας προς τρίτους, γιατί και εμείς τρίτοι είμαστε, έχει και ένα πολιτικό τίμημα. Γι' αυτό ε, εμφανίζουν μια προθυμία η δομή, ε, στη δομή τους οι διεθνείς οργανισμοί. Να σας δώσω ένα στιγμιότυπο, μια φωτογραφία αυτού που προσπαθούμε να κάνουμε τα κονδύλια που διοχετεύονται μέσα των Ηνωμένων Εθνών προσπαθούμε και διαπιστώνουμε ότι την περίοδο 2003-2006 αυξήθηκαν ε, με ταχύς ε, ρυθμούς. Την περασμένη τετραετία ενισχύθηκαν οι έλεγχοι σε πολλούς τομείς για να βεβαιωνόμαστε πάντα ότι γίνεται καλή και χρηστή διαχείριση και επιτόπου να συνεργάζονται οι υπάλληλοι του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. για να έχουμε ικανοποιητικές ε, διασφαλίσεις ότι γίνεται σωστή η διαχείριση. Οι επικεφαλείς των αντιπροσωπιών μας ε, καλούνται πλέον να αναφέρουν τακτικά στα πλαίσια των συνήθων ε, δραστηριοτήτων τους για τη συνεργασία με τους οργανισμούς. Επίσης, συμφωνήσαμε με τον ΟΗΕ να έχουμε κοινού κανόνες για προβολή και ορατότητα και διαφάνεια, έτσι ώστε να φαίνεται τι κάνουμε. Οι σημαντικοί αυτοί κανόνες ε, επίσης συνδέονται με την ε, οικονομική λογοδοσία των Ηνωμένων Εθνών. Πριν στείλουμε κονδύλια σε οποιοδήποτε διεθνή οργανισμό για να τη διχειριστεί, ελέγχουμε τον τρόπο με τον οποίο τηρούν τα στοιχεία τους, κάνουν εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους και προχωρούν στη σύναψη συμβάσεων. Έχουμε Επίσης και το δικαίωμα επιτόπου να κάνουμε ελέγχους για να διαπιστώνουμε κατά πόσο έχει γίνει σωστή διαχείριση σύμφωνα με τους κανόνες. Και φέτος τον Απρίλιο ε, ε εγκρίναμε και κανόνες ακριβώ για τη λειτουργία αυτών των ε, διερευνητικών αποστολών. Σε συνεργασία λοιπόν με τα Ηνωμένα Έθνη ε, παρακολουθούμε και αναφέρουμε για τις δράσεις για να δούμε ότι τα χρήματά μας πιάνουν τόπο. Όχι απλώς να διαπιστώνουμε ότι έγινε ένα έργο και η δαπάνη ήταν τάδε. Υπάρχουν διάφορα ιδρύματα, ταμεία και ιδιαίτερα στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν όπου δημιουργήσαμε και ειδική σελίδα γι' αυτό. Επίσης ήθελα να προσθέσω ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι για παράδειγμα στο Αφγανιστάν αλλά και στο Ιράκ Έχουμε τέτοια ταμεία, ιδρύματα, trust funds, ακριβώς επειδή δεν μπορούμε μόνοι μας να διαχειριστούμε αυτή τη βοήθεια. Δεδομένης της τόσο δύσκολης πολιτικής κατάστασης και του στρατιωτικού περιβάλλοντος που επικρατεί στις περιοχές αυτές. Ο κύριος Λιμπεράτσκι ρώτησε κατά πόσο θα συνεχιστεί αυτή η γραμμή βελτιώσεων και μας που ε, βελτίωσαμε κατά 40% πέρυσι τις επιδόσεις μας. Επίσης ρωτήσατε αν ε, αναμένεται και του χρόνου τέτοια βελτίωση. Πιστεύω πως ναι, γιατί κανονικά οι πιο δύσκολες ε, αλλαγές γίνονται στην αρχή και το 100% δεν είναι 40% συν 40 συν 20. Δεν πάει έτσι, δεν είναι τόσο απλό σε πολιτικό επίπεδο. Απαντώ τώρα στην κυρία Αγιάλα. Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση που έκανε για τους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων που θα επικρατήσουν στο μέλλον. Είναι υποσυζήτηση είναι αυτό ακόμα. Καταλήγω δε στο συμπέρασμα ότι δεν έχουν όλη την ίδια αντίληψη για αυτό το θέμα και σύμνοια. Επιτρέψτε μου να σας αναφέρω την προσωπική μου άποψη με την εμπειρία που έχω 4-5 μηνών και όχι παραπάνω, αλλά στο παρελθόν είχα κάποια διεθνή εμπειρία. Παρατηρείτε τώρα εξής η κατάσταση. Έχουμε μια κάθετη, ε, ε, ένα κάθετο διαχωρισμό ε, και Νότια Αφρική και Κούβα, όπου ο επίτροπο Ανάπτυξης είναι αρμόδιος για την αναπτυξιακή βοήθεια, την ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά και τις πολιτικές αποφάσεις και τις πολιτικές δράσεις. Η κυρία Πενίντα Φεραίρο Βάλτνερ είναι αρμόδια για το υπόλοιπο του κόσμου και για την αναπτυξιακή βοήθεια. Αλλά ο υπόλοιπο κόσμο είναι μικρό τμήμα, γιατί κυριαρχούν οι χώρε ΑΚΕ. Αυτή είναι λοιπόν η διαίρεση που έχουμε, η κάθετη ως προς τις αρμοδιότητές μας. Τώρα, με την ίδρυση της υπηρεσίας ε, ε, εξωτερικής δράσης έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να περάσουμε προς μια οριζόντια διαίρεση. Είναι μεγάλη αλλαγή και θα χρειαστεί μάλλον πολύ χρόνο. αν κοιτάξετε ένα ρολόι για να πας από το, ε, η βελόνα από το κάθε το άξονο στον οριζόντιο χρειάζεται να γυρίσει 90 μοίρες. Οπότε θα χρειαστεί και κάποιος χρόνος για να γίνει αυτή η αλλαγή και η μετάβαση. Και πού θα γίνει αυτή η εγκάρσια λοιπόν γεωγραφικά ε, γραμμή. Θα έλεγα εξωτερική δράση, η υπηρεσία αυτή εξωτερικής δράσης να αναλάβει τα στρατηγικά έγγραφα για τις χώρες, βεβαίως ε, με τη βοήθεια των υπηρεσιών ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μάλιστα σημαντική συνεισφορά. Σε ό,τι αφορά τώρα το σχεδιασμό και την εφαρμογή, την υλοποίηση των προγραμμάτων, είναι ζωτική σημασία να παραμείνει αυτό στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να μην ασχολείται μόνο με το βραχυπρόθεσμο αλλά και με το μακροπρόθεσμο σχεδιασμό ε, βάσει των ε, γράφων στρατηγικής, των εκθέσεων στρατηγικής για τις διάφορες χώρες. Αυτή είναι, η επαναλαμβάνω, προσωπική μου αίσθηση. Στην πράξη, στην αρχή, αν μη τι άλλο, επί τόπου θα παραμείνουν διαφορές μεταξύ των χωρών ΑΚΕ και των υπολείπων. Είναι προφανές αυτό. Ε, ωστόσο, θα πρέπει σιγά-σιγά να σκεφτόμαστε με τρόπο πολύ σαφή και διαρθρωμένο. Επαναλαμβάνω, βάσει της μικρής μου εμπειρίας, αυτή είναι η κεντρική ιδέα για μένα. Σε ό,τι αφορά τώρα τη μακροοικονομική βοήθεια. Σωστά είπατε, κυρία Γιάλα, ότι μπορεί να αλλάξει η κατάσταση σε μια χώρα από τη στιγμή που παίρνει κανείς μια απόφαση μέχρι να γίνει η εκταμίευση αυτή καθ' ε, είναι γεγονός. Το περιβάλλον στις χώρες αυτές είναι πάρα πολύ ρευστό και τα πράγματα δεν βελτιώνονται πάντα, καμιά φορά δυσκολεύουν. Ιστορικά δεν ήμουν τόσο πολύ υπέρ της μακροοικονομικής βοήθειας εγώ, αλλά διαπίστωσα ότι ιδιαίτερα για ένα οργανισμό όπως είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν υπάρχουν και πάρα πολλές εναλλακτικέ λύσεις. Παρόλο που είναι πάνω από 40% ε, η χρηματοοικονομική στήριξη στους προϋπολογισμούς παίρνουμε αιτήσει της τάξης των 40.000 με 50.000 που είναι πάρα πολύ μεγάλος όγκος ε, ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να ε, αναλάβουν περισσότερες ευθύνες οι αναπτυσσόμενες χώρες αν αποδεικνύουν ότι δεν είναι σε θέση να αναλάβουν την ευθύνη αυτή νομίζω πρέπει να έχουμε το πολιτικό θάρρος και το πολιτικό σθένος να παίρνουμε εμείς αποφάσεις και να λέμε ότι κοιτάξτε τέρμα η βοήθεια και πηγαίνετε να εξηγήσετε στο λαό σας γιατί σταματήσαμε να σας βοηθούμε. Λοιπόν, μαζί με την μακροοικονομική βοήθεια και, και τα αυξημένα κονδύλια που ουραίουν προς την κατεύθυνση αυτή, θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη συνειδητοποίηση. Να αναλαμβάνει ο καθένας τις ευθύνες του και καμιά φορά μπορούμε να καταλήγουμε και στην απόφαση ότι τερματίζεται η βοήθεια. Ξέρω ότι ακούγονται διάφορες ιδέες για κατηγοριοποίηση των απτυσσομένων χωρών. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα για πολλούς λόγους. Πρώτον, πολιτικά είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Αν θα πρέπει τώρα να αρχίσουμε να ταξινομούμε χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε, πολιτικά αυτό είναι πάρα πολύ λεπτό θέμα. Ε, δεύτερον, όπως πολύ σωστά λέτε, αλλάζουν οι καταστάσεις και πολύ γρήγορα. Τι θα κάνουμε εμείς, δηλαδή συνέχεια θα αναθεωρούμε την κατάταξη κάθε χώρα ή κάθε χρόνο. Και τρίτο, αν ήμουν επίτροπος ανάπτυξης εγώ, θα είχα πολύ μεγάλη ε, επιφύλαξη ως προς αυτό. Ε, κάποιος θα πρέπει να λάβει πολιτική ευθύνη για ε, ένα θέμα που δεν μπορεί 100% να το αξιολογεί και αυτό στην πολιτική θα πρέπει να το αποφεύγουμε. E- ευχαριστώ. Παρακαλώ όλοι να κρατιάστε μέσα στον ευρωπαϊκό χρόνο. Κύριε Στάς. Ο κύριος Στάς, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος γιατί είναι πολλοί ομιλητές και ο χρόνος περιορισμένος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο για τις απαντήσεις και τις υπηρεσίες του. Ε, το ερωτηματολόγιο έχει διανεμηθεί σε ό,τι αφορά την έκθεση και του κυρίου Λιμπεράτσκι και την έκθεση κυρία Αγιάλα για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Με πολύ μεγάλη προσοχή διάβασα τις απαντήσεις. Ήταν πολύ υψηλής ποιότητας. Σωστά είπε η κυρία Γιάλα ότι είναι λίγο περίεργη η κατάσταση, λίγο μυστήρια και παράξενη. Έχουμε εδώ ενωπιό μας τον Γκάριλ Τεχιούχτ που μόλις ανέλαβε πριν από τέσσερις μήνες ε, το χαρτοφυλάκιο αυτό και τώρα θα πρέπει να έρθει να λογοδοτήσει για τον προκάτοχό του. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και το εκτιμώ πάρα πολύ το γεγονός αυτό. Γιατί ο Καρλ Χόχτ παίζει εδώ πολιτικό ρόλο. Δηλαδή, η απαλλαγή δεν είναι απλώς ε, μια λογιστική άσκηση, είναι και πολιτική άσκηση. Και από την τετράμινη λοιπόν πείρα του νομίζω μπορούμε να αντλήσουμε και εμείς διδάγματα και για το πώς θα κάνουμε τις απαλλαγές στο μέλλον. Με πολύ μεγάλο λοιπόν ενδιαφέρον και προσοχή άκουσα τα όσα είπε και στο Συμβούλιο για την καλή αναπτυξιακή βοήθεια και πώς μπορεί αυτή να οργανωθεί καλύτερα με σημεία κλειδιά. Δηλαδή λιγότερα έργα να χρηματοδοτούμε, καλύτερο συντονισμό να έχουμε μεταξύ των όσων πράττουν τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ δεν μας είπατε πολύ ε, αναλυτικά πώς θα το οργανώσετε. Αν θέλετε να μας το συγκεκριμενοποιήσετε αυτό, κύριε Τεχιούχτη, σας παρακαλώ. Απαντώντας στην κυρία Γιάλα, Σέντερ, μιλήσατε για τη μακροοικονομική βοήθεια, αλλά εγώ έχω την εξής ερώτηση. Εσείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πώς οργανώνετε τον έλεγχο όταν ενισχύεται τον προϋπολογισμό μιας χώρας. Εντάξει, ας πούμε ότι αλλάζει η πολιτική κατάσταση σε μια χώρα και μπορούμε να αποφασίσουμε ότι έχει επιδεινωθεί πάρα πολύ και θα πρέπει να πάρουμε πολιτικές αποφάσεις γιατί πάνε χάλια τα πράγματα. Αλλά πώς οργανώνετε εσείς το λογιστικό και το οικονομικό έλεγχο. Και τελευταία ερώτηση. Φέτος έκανε το ελεκτικό συνέδριο ειδική έκθεση για τους λεγόμενους μη κρατικούς φορείς, non-state actors. Τι είναι αυτή και πώς ε, δίνεται αναπτυξιακή βοήθεια εκεί. Γιατί η μακροοικονομική απευθύνεται στα κράτη. Και ποια είναι η σχέση τους εκεί και ο ρόλος των Ηνωμένων Εθνών, εντάξει απαντήσατε, έτσι κι αλλιώς του χρόνου θα το δούμε αυτό στην απαλλαγή γιατί εξ όσων κατάλαβα το ελεγκτικό συνέδριο θα κάνει ειδική έκθεση του Κάιλ Πίνγκστεν για τα Ηνωμένα Έθνη οπότε με μεγάλο ενδιαφέρον θα τα συζητήσουμε και θα τα συμπεριλάβουμε στις εργασίες μα αυτά του χρόνου. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, κύριος Επίτροπος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με τα κράτη-μέλη πρώτον, δεν μπορώ να πω σε λεπτομέρειες, δεν έχουμε το χρόνο, αλλά αυτό που διαπιστώνετε εσείς τι είναι. Ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά κυρίως τα κράτη-μέλη, έχουν πάρα πολλές χώρες με τις οποίες συνεργάζονται και πολλούς τομείς στο εσωτερικό των κρατών αυτών. Και το σύνολο, το άθροισμα οδηγεί σε πάρα πολύ ε, διαφορετικούς τομείς, κλάδους που θα πρέπει να συμφιλιώνονται μεταξύ του. Ωστόσο, αυτό που θα έπρεπε να κάνουν ε, οι υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το υποστηρίζω προσωπικά είναι να προσπαθήσουμε να έχουμε κάποιες χώρες δωρητές, περιορισμένο αριθμό. Δηλαδή τα κράτη-μέλη της Ένωσης μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κοιτάμε ένα περιορισμένο ε, αριθμό δικαιούχων κρατών και περιορισμένους τομείς. Ας πούμε να φτιάξουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα και να δούμε ποια είναι η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των προγραμμάτων και πώς μπορούμε να λειτουργούμε καλύτερα. Έχω καταλάβει ότι ορισμένα κράτη-μέλη είναι πρόθυμα να κάνουν ένα τέτοιο πιλωτικό πρόγραμμα. Έκλεισε το μικρόφωνο δυστυχώς του Μίλτου. Μετά από τέσσερις μήνες ούτε ένα μικρόφωνο μπορώ να ανοίξω. It simply fell out, Απλώς κατέρευσε το μικρόφωνο. Έλεγα λοιπόν ότι ορισμένες χώρες εμφανίζουν την προθυμία αυτή να κάνουν πολιτικό πρόγραμμα και να το κάνουμε. Όταν έχουμε 27 χώρες που κάνουν μια συμφωνία με μια χώρα, ε, του χρόνου να προσπαθήσουμε να στήσουμε ένα σοβαρό πιλωτικό πρόγραμμα. Τώρα, για τη μακροοικονομική βοήθεια. Πώς την ελέγχεις. Κοιτάξτε. Αυτό εξαρτάται πάρα πολύ από τις επιτόπου υπηρεσίες μας, τις αντιπροσωπίες μας δηλαδή. Μου έκανε εντύπωση και στην προηγούμενη ιδιότητά μου πόσα πράγματα γνωρίζουν οι άνθρωποι που είναι εκεί οι δικοί μας για την κατάσταση επιτόπου και καταφέρνουν όχι να μιλάνε έτσι γενικόλογα, αλλά να γνωρίζουν ποιε είναι οι αδυναμίες, πού χωλαίνει ένας οργανισμός. Όταν πας σε μία οργάνωση από μακριά να τη βλέπεις, σου φαίνεται πάρα πολύ οργανωμένη και διαρθρωμένη, αλλά όσο πλησιάζεις τόσο αρχίζεις και βλέπεις τις αδυναμίες και τα κενά. Αυτά τα γνωρίζουν οι δικοί μας άνθρωποι εκεί και μπορούν να μας βοηθούν ε, τη δημιουργία των θεσμών, όπως λέγεται, αυτό, institution building και στις διάφορες επίσης ε, λογιστικές ε, δράσεις και λογιστικούς ελέγχους. Δηλαδή, να δούμε πού μπορούμε και σε ποιο επίπεδο δίνουμε ε, μακροοικονομική βοήθεια. Αν μπορεί να γίνει σε περιφερειακό επίπεδο, σε τοπικό επίπεδο, επίπεδο επαρχίας, αυτό εξαρτάται από την οργάνωση της κάθε χώρας. Να μην είναι πάντα κεντρική βοήθεια, αλλά να πηγαίνει όσο γίνεται πιο κοντά στον πολίτη, ε, στον τελικό δικαιούχο, να εφαρμόζουμε την επικουρικότητα. Οι μη κρατικοι φορει φορείς, non-state actors, Εργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό το τομέα. Είναι πάρα πολύ περίπλοκο αλλά και αναγκαίο ε, γιατί από τη μια ε, συνεργαζόμαστε με κράτη αλλά και με μη κρατικού φορεί που μπορεί να είναι μη κυβερνητικέ οργανώσει, για παράδειγμα. Και είναι πολύ σημαντικό στοιχείο και πολύ σημαντικό πολιτικό στοιχείο στο εσωτερικό των κρατών μελών. Θα πρέπει να το λαμβάνει υπόψη αυτό και ε, η κυβέρνηση. Πολλές ε, χώρες δίνουν μεγάλη σημασία στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και θα πρέπει να έχουμε ένα συγκεκριμένο επίπεδο εκεί. Γενικά λοιπόν υπάρχει μια αρχή που λέγει ότι οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις είναι σημαντικές για μια χώρα και λιγότερο σημαντικές για μια άλλη. Ε, ξέρουμε ότι σε χώρες που καταραίουν ή έχουν καταρρεύσει είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση των μη κυβερνητικών οργανώσεων ε, αλλά αν δεν υπήρχαν δεν θα μπορούσαμε να είχαμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία, τη βασική κάλυψη του πληθυσμού. Αλλά ε, έχει σημασία να υπάρχει ένας πολιτικός διάλογος και επίσης να ε, πηγαίνουμε και σε μεγαλύτερε μη κυβερνητικέ οργανώσει. Ξέρω ότι είναι πολύ συμπαθέ και ακούγεται ευχάριστο να συνεργαζόμαστε με μικρέ μη κυβερνητικέ οργανώσει, αλλά με τι μεγαλύτερε είναι πιο αποτελεσματικό, έχει και πιο διαρθρωμένο διάλογο και μεγαλύτερο αντίκτυπο στον προγραμματισμό. Τώρα έρχονται όλα τα προγράμματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεκάδες χιλιάδες ε, μικρές ΜΚΟ, αλλά καλύτερα είναι μεγαλύτερες που έχουν μια συγκεκριμένη αποστολή, έχουν μια οργάνωση, μια διάρθρωση, μπορούν να μπουν από τη φάση του σχεδιασμού και του προγραμματισμού και να έχουν μεγαλύτερη συνεισφορά. Άλλοι τέσσερι θέλουν να μιλήσουν. 10 ε. και τέταρτο θα διακόψουμε το σημείο αυτό για να προλάβουμε και τα υπόλοιπα. Γκρέσλε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι τμήμα της λύσης εγώ. Κύριε Πίτροπε, εγώ να σας πιστέψω για τη μακροοικονομική βοήθεια. Όταν λέτε ότι όποιος δεν διαχειρίζεται καλά, τέρμα τα λεφτά. Ωραία, ποια καταγγείλατε το 2008 και 2009 μακροοικονομική βοήθεια. Εάν το 2008 δεν υπήρχε τέτοια καταγγελία και διακόπη. Σε σχέση με αυτό μπορώ να σας μιλήσω για την Κένια δύο ή τρεις ημέρες πριν τις βουλευτικές εκλογές πήρε 40 εκατομμύρια ευρώ ή δολάρια, δεν θυμάμαι η Κένια και δεν φαίνεται να ψάχνει πάρα πολύ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, πρώτον, ποια βοήθεια κόψατε και δεύτερη, πώς αποκλείεται την κατεπανάληψη ε, λάθος διαχείριση από την Κένια, ας πούμε. Άλλη ερώτηση αφορά μια ειδική οργάνωση της αναπτυξιακής βοήθειας, γιατί εκεί συμμετέχουν πολύ ε, διαφερόμενοι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πολλές γενικές διευθύνσει. Τώρα με τι της Λισαβόνα είναι χειρότερα για μας τα πράγματα, γιατί δεν καταλαβαίνουμε πραγματικά ποιο θα είναι αρμόδιος για τι πράγμα. Οπότε θα είχα κάποια πράγματα να ζητήσω από την επόμενη οργάνωση, μια παράκληση ή πολλέ παρακλήσει. Περιμένουμε σαφή διαχωρισμό από τη διπλωματική υπηρεσία. Η αναπτυξιακή βοήθεια θα παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έπεσε το μικρόφωνο και της κυρίας Γκρέσ. Εμείς αναμένουμε ε, ε, οι ε, επιτόπου στις αντιπροσωπείες υπαλλήλοι να είναι της αναπτυξιακής βοήθειας της αρμόδιας γενικής διεύθυνσης. Ε, μην γίνει το μεγάλο μπέρδεμα τώρα στην εξωτερική ε, υπηρεσία. Θα πρέπει να υπάρχει και μια σταθερότητα. Να επανέλθω σε μια στατιστική που πήραμε με τώρα στην Επιτροπή Ελέγχου και ε, αφορά το προσωπικό των αντιπροσωπιών. 186% ε, αύξηση έχουμε από το 2000. Είναι πάνω από 5.000 οι εργαζόμενοι ε, και η μισή και παραπάνω είναι ντόπιοι στην κάθε χώρα. Επιτρέπετε να σας ερωτήσω πόσοι σε κάθε αντιπροσωπεία ασχολούνται με την άπτυξη και βοήθεια. Ξέρω ότι ίσως να μην είστε σε θέση να μου απαντήσετε τώρα. Αλλά πόσοι εργαζόμενοι στις αντιπροσωπείες αυτές έχουν επιφορτιστεί με την αναπτυξιακή βοήθεια. Και θα ήταν χρήσιμο επίσης να μάθουμε και για τις Βρυξέλλες. Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξη, Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακή Βοήθεια. Πόσοι από τους υπαλλήλους αυτούς ασχολούνται με την αναπτυξιακή βοήθεια. Καταλαβαίνετε που το πάω για να καταλάβουμε τι θα παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι θα πάει στη διπλωματική υπηρεσία. Ευτυχώ δεν σα χάνουμε από επίτροπο και χαίρομαι γι' αυτό και θα ήθελα οι αρμόδιοι επιτροποί στη Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμμετέχουν περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν γιατί βλέπουμε ήδη κάποια κομμάτια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεπουλάνε, να εκποιούν διάφορε υπηρεσίε χωρί να ρωτηθούν καν οι ενδιαφερόμενοι. Και για τη διεθνή οργάνωση αυτό δεν βοηθάει και θα, θα λουστούμε εμείς μετά. Και θα ερχόμαστε να λύνουμε τα προβλήματα με σύγκρουση αρμοδιοτήτων σε επιτροπές του Κοινοβουλίου. Άλλη ερώτηση για τον ΟΗΕ. Με τον προηγούμενο πρόεδρο της Επιτροπής μας κάναμε πολύ ωραίο ταξίδι στον ΟΗΕ και είδαμε στο κουσιφοπέδιο ότι ο ΟΗΕ δεν διαχειρίζεται πάντα καλά τα χρήματά μας στο Κωσυφοπέδιο ο ΙΕ ΕΕ είναι τμήμα του προβλήματος και όχι τμήμα της λύσης και υποθέτω συμβαίνει και αλλού αυτό. Πώς παίρνετε εσείς την απόφαση ε, να διαχειρίζετε τα κονδύλια αυτά ο ΙΕ και όχι εμείς, εσείς δηλαδή. Και επίσης πόσα κονδύλια ε, διατέθηκαν το 2008 και γραπτός παρακαλώ στον ΟΗΕ για να τα διαχειριστεί δικά μας αναπτυξιακά κονδύλια. Ευχαριστώ. Επειδή οι ερωτήσεις είναι πολύ συγκεκριμένες, ίσως να μην εξαντληθούν στην προφορική απάντηση, θα μπορεί η Κομισιόν να απαντήσει γραπτά, αν θέλει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Γκρέσλε, Ρωτήσατε πού δαπανήθηκε η υποστήριξη του προπολογισμού. Δεν έχω μαζί μου τον κατάλογο. Από ό,τι ξέρω, ε, που, που διακόπη προσωρινά. Μόνο σε μία χώρα διακόπη, στη Μαδαγασκάρη, μετά ένα πραξικόπημα. Εκεί διακόπη. Είχαμε διακοπές και το 2009, αυτό όμως αφορά το επόμενο έτος. Βέβαια και ορισμένε άλλε χώρε επλήγησαν από την χρηματοπιστωτική κρίση. Και αυτό δημιούργησε καθυστερήσεις. Πάντως αυτό δεν εκτροχίασε την υποστήριξη του προϋπολογισμού το 2008 με εξαίρεση τη Μαδαγασκάρη. Αναφερθήκατε στην Κένια. Λίγες μέρες μετά τις εκλογές εδόθησαν 40 εκατομμύρια. Τα χρήματα υπήρχαν και πριν τις εκλογές. Δόθηκαν λίγες μέρες μετά, στις 27 Δεκεμβρίου αν θυμάμαι καλά, επειδή ήταν τέλος της χρονιάς. Για την Κένια κανένας δεν περίμενε ξαφνικά μετά τις εκλογές να έχουμε αυτή τη φοβερή αντιπαράθεση, σύγκρουση με εθνοτική διάσταση. Η Κένια θεωρείται μια από τις πιο σταθερές χώρες της Αφρικής. Για να καταλάβετε τι σημαίνει η σταθερότητα στην Αφρική. Ξαφνικά δηλαδή μπορεί να ξεσπάσει μια σύγκρουση ως τυφώνας. Και είναι εύκολο να λέμε ναι, έπρεπε να περιμένετε, να δείτε αν θα συμβεί κάτι τέτοιο μετά τις εκλογές. Δεν το περιμέναμε. Για τη Λισαβόνα και τις επιπτώσεις απάντησα ήδη. Σε ερώτηση της κυρίας Αγιάλα. αντιπροσωπείες το προσωπικό. 2.300 άτομα δουλεύουν σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι όλοι προσωπικό της Κομισιόν. Οι υπάλληλοι είναι και ντόπια στελέχη. 2.300. τρακόσι. Κόσοβο. Δεν την ξέρω την έκθεση, έχω πάει κάποιες φορές στο Κόσοβο. Δεν είναι εύκολη περιοχή για να εφαρμόσει κανείς προγράμματα. Και αν δείτε και το Αφγανιστάν, θα έλεγα ότι μπορεί να έχετε πιο ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Και μην επικρίνετε τα άτομα που δουλεύουν κατά από δύσκολες συνθήκες. όλα αυτά τα προγράμματα είναι σχετικά σε περιοχές όπου υφίστανται σειράξεις. ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω για να συγχαρώ ειλικρινά από την ε, Ολλανδία για το διορισμό του στη νέα θέση στην επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να το ευχηθώ κάθε επιτυχία. Θα ήθελα όμως να επανέλθω στα σημερινά και την αναπτυξιακή βοήθεια και την ανθρωπιστική βοήθεια. Στην αρχή μας είπατε κύριε Επίτροπε ότι θα πρέπει να είναι αποτελεσματική και με καλή διαχείριση και διαφανής η βοήθεια. Αυτό είπατε εισαγωγικά. Και μετά μας λέτε ε, πού είναι η αποτελεσματική βοήθεια. Κατά την άποψή μου θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν γιατί είναι περιορισμένα τα κονδύλια για την εξωτερική πολιτική και επανέρχομαι στη γενική μακροοικονομική βοήθεια. Τα είπαν οι προλαλήσαντες να εμφαθύνω λίγο περισσότερο στη συνοχή Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα κράτη-μέλη. Πώς είναι δυνατόν, αν θέλετε να είστε αποτελεσματικοί, να υπάρχουν κράτη-μέλη που σταματούν τη μακροοικονομική βοήθεια Άλλα προγράμματα συνεχίζουν, αλλά δεν δίνουν άμεσα μακροοικονομική βοήθεια λόγω του καθεστώτος ε, κάπου. Ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δίνει μακροοικονομική βοήθεια αμέσω μετά, μόλις σταματήσουν τα κράτη-μέλη. Πού είναι το νόημα και η ανοησία της γενικής μακροοικονομικής βοήθειας εδώ. Παράδειγμα, το Νοέμβριο του 2008 λέει η Ολλανδία. Στη Ρουάντα, στην Ουγγάντα, συγγνώμη, ε, γιατί παραβίασαν το εμπάργο των όπλων ε, στη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό. Σταματούμε τη μακροοικονομική βοήθεια, αλλά χρηματοδοτούμε άλλα μικρά προγράμματα. Την ίδια περίοδο έρχεται ο Επίτροπο κύριο Μισελ. Λυπάμαι, τώρα έρχεται να λογοδοτήσετε για πράγματα που έκαναν οι προκάτοχοί σα. Στην ίδια περίοδο έρχεται και δίνει από τα ευρωπαϊκά κονδύλια 175 εκατομμύρια. Άλλο παράδειγμα, πιο πρόσφατο, η Τανζανία τον Αύγουστο του 2009 350 εκατομμύρια ευρώ ε, μακροοικονομική βοήθεια παρόλο που διάφορα κράτη-μέλη, όχι ένα μόνο, σταματούν τη χρηματοδότηση προς την Τανζανία. Στο μεταξύ λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε καλά, δώσαμε την πρώτη δόση αλλά θα δούμε στις επόμενες τι θα κάνουμε. Σπιράλ, ε, κλιμακώνεται. Ε, θα το λάβουμε υπόψη την επόμενη φορά, την επόμενη δόση των 305 εκατομμυρίων. Τώρα αυτή τη στιγμή τι γίνεται, πώς έχει κατάσταση. Γιατί το θέμα είναι να εξασφαλίζετε την αποτελεσματικότητα και τη συνέχεια και τη συνέπεια. Πέρα από τα πιλωτικά προγράμματα που μας αναφέρετε. Ξέρω ότι θα πείτε ότι είναι θέμα του αντικαταστάτου μου αυτού, αλλά Όποιος έχει πείρα στην πολιτική και εσείς έχετε πείρα θα μπορέσετε να δώσετε και καλές συμβουλές. Αν δεν μείνω να ακούσω την απάντησή σας, δεν είναι επειδή είμαι αγενής, με περιμένουν έξω δύο δημοσιογράφοι, αλλά οι συνεργάτες μου είναι παρόντες και θα τα σημειώσουν αυτά που θα πείτε. Yeah, uh, Ευχαριστώ. Απάντηση. Ευχαριστώ κυρία μου. Και για τα συγχαρητήρια δεν έχω συνηθίσει να με συγχαίρουν οι Ολλανδοί. Πολύ με ευχαριστεί αυτό και με χαροποιεί. Λοιπόν, τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη συνεργασία με τα κράτη-μέλη και τη συνέπεια και τη συνοχή. Ενδιαφέρουσα ερώτηση. Διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να κάνει ε, άλλη εκτίμηση να έχει άλλη κρίση για κάποια κράτη, αλλά όταν τα κράτη-μέλη διαφέρουν στην άποψή τους, ε, αυτό πλήττει και τη διεθνή εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι δεν τη βοηθάει πάρα πολύ τη διεθνή εικόνα της Ένωσης. Γιατί δεν εμφανίζουμε συνοχή προς τα έξω, σίγουρα. Και υπάρχει εξήγηση. Διατηρούμε την ανεξαρτησία μας, αλλά καλό θα ήταν να συντονίζομαστε γιατί δεν δίνουμε καλή εντύπωση. Να σας πω απαντώντας. Πρώτον, Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας οργανωμένος τρόπος διαβούλευσης μεταξύ των κρατών μελών που δραστηριοποιούνται σε μια χώρα και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έτσι ώστε ο καθένας να αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Και πριν ε, δοθεί μια βοήθεια να υπάρχει συνεννόηση. Μιλήσατε για την ε, ε, Ρουάντα, την Τανζανία, την Ικαράγουα. 10 εκατομμύρια ευρώ ε, διαθέσαμε εκεί και η δική σας χώρα και κάποιες άλλες πήραν αποφάσεις. Λοιπόν, οργανωμένη διαβούλευση γι' αυτό. Δεύτερον, σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να γίνει διάκριση μεταξύ ε, διαλόγου, πολιτικού διαλόγου και διαλόγου για επιμέρους ζητήματα πολιτικής. Δηλαδή policy dialogue και political dialogue λέγεται αυτό στα αγγλικά. Στο Κοτονού γίνεται λόγος για την επιμέρους πολιτική, αλλά ο πολιτικός διάλογος είναι στο άρθρο 8. Και εκεί μπαίνουμε σε θέματα αδίκησης κρατικής μηχανής, ελέγχου για τη μακροοικονομική βοήθεια. Αλλά δεν μπορούμε να ε, βάζουμε θέματα δημοσιονομικά και λογιστικά σε αυτά που είναι πολιτικός διάλογος. Στη Ρουάντα, ας πούμε, αυτό ήταν το θέμα με τη στάση τους στο Ανατολικό Κονγκό, όπου ξεκίνησαν μεγάλες ε, συνομιλίες. Είναι καθοδόν ε, λοιπόν, αυτή η διαδικασία χρειάζεται συντονισμός και βεβαίως θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε και να οργανωνόμαστε έτσι ώστε προς τα έξω να έχουμε μία φωνή. Αν δεν το κάνουμε αυτό, αποδυναμωνόμαστε ο μόνοι μας και δεν νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε τέτοιο στόχο. Εξαντλήθηκε ο χρόνος. Παρακαλώ τα δύο συνεδέρους που ήταν να μιλήσουν να είναι πολύ σύντομη στην ερώτηση. Ο Επίτροπος θα απαντήσει γραπτά. Ολμάγερ και μετά ο Ντί. Αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο παρά το χωριμένο της ώρας. Καταρχάς θα ήθελα να ρωτήσω κάτι για τα Ηνωμένα Έθνη έχει καν νόημα να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με τα Ηνωμένα Έθνη σε αυτή τη βάση αφού 5% του διοικητικού προϋπολογισμού καλύπτεται και από τα δικά μας κονδύλια, τα κοινοτικά και έχουν μια στάση άρνησης συνεχώς για σοβαρό συντονισμό για τα διάφορα προγράμματα επιτόπου. στο λογιστικό έλεγχο και στην τήρηση των βιβλίων δεν τηρούν καν τα ελάχιστα πρότυπα που θα περίμενε κανείς από ένα τέτοιο οργανισμό. Δεύτερον, θα ήθελα να συμφωνήσω και εγώ με την ανησυχία της κυρίας Γκρέσλε. Φοβάμαι ότι στη νέα οργάνωση ε, των διαφόρων τομέων θα έχουμε νέες θολούρες και ασάφειες και αδιαφάνειες και θα έρθουμε και στην επόμενη έκθεση να λέμε τα ίδια για περισσότερα προβλήματα. Έχω μία παράκληση λοιπόν και μία ερώτηση υπάρχει προθυμία να ενημερώνεται το Κοινοβούλιο για την ανακατανομή, το σχεδιασμό των υπηρεσιών που κάνετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τρίτον, άκουσα ότι υπάρχουν διάφορα ταμεία, ιδρύματα, trusts, ε, με τα οποία έχετε, καλή εμπειρία για την εκτέλεση των προγραμμάτων. Ότι έχει βελτιωθεί πολύ η κατάσταση σε σχέση με άλλους τομείς που έχουμε συνηθίσει. Ε, δεν θα είχε νόημα εκεί λοιπόν να ανατρέχουμε σε τέτοιους εταίρους αφού είναι επιτυχή με ένα λέτε τα, προβλημα... τα προγράμματα. Συγγνώμη. Και μια τελευταία ερώτηση. Φαίνεται να υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα εδώ στις κεντρικές υπηρεσίες της Europe Aid. Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα του προσωπικού. Μετατίθενται κάθε τρία χρόνια. Έρχεσαι τον πρώτο χρόνο, γνωρίζεις κόσμο, ένα χρόνο δουλεύεις και τον τρίτο χρόνο αρχίζεις και ε, ετοιμάζεσαι να φεύγεις και τον τέταρτο χρόνο έρχεται νέος. Δεν μπορεί να σταματήσει αυτό γιατί έχετε μεταθέσει κάθε τρία χρόνια. Euh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, ως βουλευτής εγώ έχω μπερδευτεί και επαναλαμβάνω κάτι που είπα. Η Ένωση θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τις δομές της. Κάντε μια, δώστε μια καλή απόδειξη του οριζόντιου και του κάθετου. Έχετε τρεις επιτρόπους, έχετε πολλές γενικές δευθύνσεις που ασχολούνται. Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Εμείς προτείναμε να περάσουν από τον κοινωτικό προπολογισμό όλα αυτά. Ζητήσαμε έρευνα, μελέτη. Τι έγινε με αυτό. Για την Τράπεζα Επενδύσεων, όλα τα κράτη είναι ακατανόητο. Κανεί δεν καταλαβαίνει ποιο κάνει τι, ποιο ελέγχει τι. Και η γενική αίσθηση, όχι του πολίτη, των φορέων, όταν αυτά τα διεθνή θέματα δεν ελέγχονται σωστά. Όταν μιλάμε για δημόσια κονδύλια, αυτό δεν είναι σωστό. Και υπάρχουν και χώρες όπου η διαφθορά είναι το εθνικό σπορ. Και λυπάμαι, κύριε Πρόεδρε, διότι στις ΑΚΕ στον ιστορικό κανονισμό βάλαμε όρον ότι πρέπει να είναι στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου και Ανάπτυξης στις αντιπροσωπείες γιατί πρέπει να είμαστε σε θέση να βλέπουμε επιτόπια τι συμβαίνει. Σας κάνω μια πρόταση κύριε Επίτροπε. Είπατε η Κομισιόν να μείνει το εκτελεστικό εργαλείο. Έχετε δίκιο. Αλλά όταν έχουμε τη συνθήκη της Λισαβόνας, έχουμε το θεσμικό τρίγωνο κάντε μια ε, συμμαχία με το Κοινοβούλιο. Μπορεί να φαίνεται ότι δεν αγαπάμε τις επιτρόπους. Εμείς επικυρώνουμε την εκλογή των επιτρόπων, συνεργαζόμαστε πολύ με σας και έχουμε και την ψήφο μομφής κατά της Κομισιόν που μπορεί να επηρεάσει τα πράγματα. Είδαμε τι έγινε με τον Μάντεσεν και τον Μακρύβ που έχουν επιμέρους επιρροή. Συνεργαστείτε με εμά, μην κοιτάτε μόνο του πρωθυπουργού. Ο κύριο Φαντροπόη εξηλέγει. δεν ήρθε καν να μα πει καλημέρα. Πάει και βλέπει πρωθυπουργού σε όλο τον κόσμο, δεν ήρθε στην Ολομέγεια να μα χαιρετήσει. Κάντε πολιτική συμμαχία με το κοινοβούλιο και θα κινηθούν τα πράγματα. Και στην εξωτερική αυτή δράση επιτέλου θα υπάρξει κάποια ακολουθία. Πρόεδρο, ευχαριστούμε τον Αντιπρόεδρο Αουντή που μας θύμασε τα κυριαρχικά δικαιώματα του Κοινοβουλίου. Δυστυχώς τελείωσε η ώρα για το σημείο αυτό. Η Κομισιόν και για τις τελευταίες ερωτήσεις μπορεί να στείλει γραπτές απαντήσεις και σχόλια. Ευχαριστούμε τον Επίτροπο. Καλή του μέρα. Και περνάμε στο 7. Ετήσια έκθεση της Επιτροπής Εποπτείας Όλαφ. Στον πρόεδρο Πίτερ Στρεμπέργκ. Tack så mycket, herr ehm, ordförande, för ordet. Σας παρακαλώ λίγη προσοχή, λέει ο Πρόεδρος. Παρακαλώ, κύριε Στόμπερκ. Ευχαριστώ πολύ. Αποχώρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορείτε να συνεχίσετε. Ευχαριστώ πολύ. Περίμενα απλώς ε, να αραιώσουμε λίγο εδώ. Εξ ονόματος λοιπόν της Επιτροπής Εποπτείας θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση να έρθουμε εδώ στην Επιτροπή σας να σας δώσουμε και μία εικόνα του πώς εργαζόμαστε. Ε, καταρχάς να σας συστήσω τα μέλη της Επιτροπής μας. Ε, στα δεξιά μου έχουμε τον κύριο Κάμα Γιώργη, ο οποίος ήταν επικεφαλής της εισαγγελίας στην Ουγγαρία, τώρα είναι υπεύθυνος ε, σε θέματα εφαρμογής εποπτείας. Έχουμε και τον πρώτο αντιπρόεδρο της Επιτροπής μας εδώ. Ε, ήταν ο πρώτος αντιπρόεδρος όταν ξεκινήσαμε πριν από τέσσερα χρόνια. Ήταν ε, αρμόδια σε θέματα εποπτείας στο Ηνωμένο Βασίλειο και τώρα είναι επικεφαλής ε, του, πάνελ, ε, του συμβουλευτικού πάνελ ε, κατά της απάτης. Έχουμε και άλλα δύο μέλη τα οποία δυστυχώς δεν μπορούν να είναι εδώ σήμερα. Ο Ντίτ Γιάρτου, ο οποίος είναι πρώην μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πολύ γνωστός νομίζω στην Επιτροπή σας, γιατί ήταν και πρόεδρος εδώ. Και επίσης έχουμε και τον Λούις Λόπες Σάνσα, που ήταν και αυτός πρώην πρόεδρος της Επιτροπής. Τελείωσε τη θητεία του πριν από κάποιες εβδομάδες και έδωσε τη σκητάλη σε μένα και ήταν στο το δικαστήριο της Ισπανίας. Εγώ λέγομαι Πίτερ Στρόμπερκ, μόλις ανέλαβα καθήκοντα ως ε, πρόεδρος. Πριν ήμουν διευθυντής του Εποπτικού ε, Συμβουλίου Δημοσίων Λογαριασμών στη Σουηδία. Πρόκειται για ένα φορέα ο οποίος είναι αρμόδιος ε, για ε, εσωτερικούς ελεγκτές ιδιωτικών ε, επιχειρήσεων. Όπως σας είπα λοιπόν, είμαι φρέσκος φρέσκος σε αυτή τη δουλειά και στην Επιτροπή μας απλά ανταλλάξαμε ρόλους. Δεν είναι τα πράγματα όπως σε άλλα όργανα όπου έχουμε μια περιτροπή προεδρία από τη Σουηδική στην Ισπανική. Εμεί θα τα κάναμε ανάπαδα. Αλλάξαμε από την Ισπανική στη Σουηδική Προεδρία στην Επιτροπή μα γιατί μα αρέσει να είμαστε ανεξάρτητοι. Να σα δώσω λίγο μια εικόνα του πώ εργαζόμαστε και θα εστιάσω σε λίγα σημεία. Ε, τι ακριβώ κάνουμε στην Επιτροπή, ποια είναι τα καθήκοντά μα, τι θέλουμε να επιτύχουμε, τι κάναμε πέρσι στην ετήσια έκθεση και να δώσουμε και μία συνοπτική εικόνα γι' αυτό και να δούμε και τι γίνεται με το ερευνητικό έργο της Όλαφ. Κατόπιν φυσικά είμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια και συζήτηση. Η Επιτροπή Εποπτείας έχει ως πιο σημαντικό καθήκον τον τακτικό έλεγχο των ερευνητικών δραστηριοτήτων της Όλαφ θέλει να υποστηρίζει και να διαπιστώνει τι γίνεται στο δικαστήριο, να καθορίζει την ανεξαρτησία της μέσω τακτικών ελέγχων και επειδή η Όλαφ είναι υποχρεωμένη να μας υποβάλει εκθέσεις ως ε, ε, Επιτροπή Εποπτείας, λαμβάνουμε σχετική τεκμηρίωση, λαμβάνουμε πληροφορίες, η Όλαφ πρέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα να ε, μας δίνει μια εικόνα του τι γίνεται με τις ε, επιθεωρήσεις τους ε, και τι διαπιστώνει και αν μια διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί εντός εννέα μηνών από τη στιγμή που ξεκίνησε και αυτό θα πρέπει να μας το αναφέρει με κάποια ε, σχετική αιτιολόγηση για το γιατί καθυστέρησε. Επιπλέον, η Όλαφ θα πρέπει να αναφέρει στην Επιτροπή Επιοπτείας αν οποιοδήποτε όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, υπηρεσία, οργανισμός δεν έχει λάβει τα μέτρα τα οποία έχει συστήσει η Όλαφ ε, κατά τους ελέγχους της και επίσης η Όλαφ θα πρέπει να μας αναφέρει πότε διαβιβάζει μία έρευνα σε ένα ε, ερευνητικό φορέα του κράτους μέλους. Επίσης, πρέπει να εξετάζουμε και τις διάφορες πτυχές του τι ακριβώς κάνει ΟΛΑΦ κατά τις έρευνές της και να ε, διαβάσουμε πληροφορίες και σε άλλους οργανισμούς. Το έχουμε κάνει ε, επανειλημμένος, για παράδειγμα στην έκθεση The Minimis, στην οποία θα αναφερθούμε και εντός ολίγου. Έχουμε και κάποια άλλα στοιχεία τα οποία προέκυψαν λόγω ε, ερευνών οι οποίες ε, δεν κατέληξαν σε κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα και εκεί κοιτάμε να δούμε τι γίνεται. Και έχουμε και κάποια προγράμματα τα οποία εξεργοζόμαστε αυτή τη στιγμή και θα συνεχίσουμε να έχουμε εκθέσεις γι' αυτό. Θα έχουμε ξεχωριστές εκθέσεις οι οποίες βέβαια θα συμπεριληφθούν στην ετήσια έκθεση. Όπως σας είπα λοιπόν έχουμε μία ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητές μας και η Επιτροπή πρέπει επίσης να εκφράσει και την άποψή της για τον προτινόμενο προπολογισμό της Όλαφ. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς εμείς ως Επιτροπή Εποπτείας διεξάγουμε τα καθήκοντά μας, πώς τα βλέπουμε, ποια θεωρούμε ότι είναι οι πιο σημαντικές ε, πτυχές κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μας. Το πιο σημαντικό, και αυτό νομίζω προκύπτει από τους κανονισμούς, είναι να διασφαλίσουμε ότι η ερευνητική ε, διαδικασία γίνεται με το σωστό τρόπο, ε, είναι συνεχής και δεν υπάρχουν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. Και κατά πόσον η ε, όλα ασχολείται με αυτά που είναι σημαντικά. Αν θέτει δηλαδή προτεραιότητες βάσει αυτών που ενδιαφέρουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να γίνει αυτή η εποπτική δουλειά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Όλαφ έχει μια στρατηγική την οποία την έχει σκεφτεί καλά, είναι παγιωμένη και την εφαρμόζει και σωστά. Πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι η Όλαφ διεξάγει τα καθήκοντά τους με καλά θεμελιωμένες μεθόδους. Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που εξετάζουμε και επίσης θεωρούμε ότι δουλειά μας είναι να παρακολουθούμε και τι κάνει η Όλαφ, δηλαδή να διασφαλίσουμε ότι οι έρευνες γίνονται ε, αμερόλεπτα, αποτελεσματικά και ότι υπάρχουν τακτικοί έλεγχοι με τους επικεφαλείς της ε, Όλαφ, ε, τα διάφορα τμήματα και τους εμπειρογνώμονες, καθώς επίσης και τη διεύθυνση φυσικά, για να είμαστε βέβαιοι ότι γίνεται κατάλληλη ανταλλαγή απόψεων και μπορούμε να συζητήσουμε τα ερευνητικά τους καθήκοντα. Για να γίνουν όλα αυτά και να έχουμε μία εικόνα για το κατά πόσον η έρευνα διεξάγεται χωρίς να υπάρχει επιρροή από εξωτερικούς παράγοντες. Ε, έτσι, εποπτεύουμε την ανεξαρτησία της Όλαφ κατά τις ερευνητικές της δραστηριότητες. Αυτό είναι το βασικό καθήκον που μας έχουν αναθέσει τα τρία θεσμικά όργανα. Αυτό λοιπόν που χρειαζόμαστε για να διεξάγουμε τα καθήκοντά μας, ε, για να έχουμε πρόσβαση σε υλικό από την Όλαφ για παράδειγμα, ε, συμπεριλαμβανομένης και το εις βάσης δεδομένων, ε, δεδομένων της. Θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση σε όλους τους εργαζομένους της Όλαφ. Γι' αυτό και εμείς χρειαζόμαστε κατάλληλο γραμματιακό προσωπικό. Να σας πω ότι τα έχουμε όλα αυτά. Έχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειαζόμαστε. Έχουμε πρόσβαση στα αρχεία που χρειαζόμαστε και εδώ να επισημάνω ότι και το προσωπικό της Όλαφ σε όλα τα επίπεδα ε, μας μιλάει πάντα με ιδιαίτερη χαρά. Ποτέ δεν θεωρήσαμε ότι πρέπει να πιέσουμε κάποιον για να μας ε, απαντήσει και θεωρούμε λοιπόν ότι η συνεργασία με την Όλαφ είναι εξαιρετική και οι επαφές με την Τροπή Εποπτείας είναι εξαιρετικές. Μας δίνεται δε η εντύπωση ότι η Όλαφ μας ακούει και συνήθως ε, προσπαθεί να προσαρμοστεί στις συστάσεις μας. Φυσικά υπάρχουν ε, ε, περιπτώσεις οι οποίες ερίζουν οι απόψεις, ε, κάπου ε, τα πράγματα δεν έχουν πάντα ολοκληρωθεί, αλλά γενικά η Όλαφ τίνει να έχει μια πολύ θετική εικόνα για τα όσα έχουμε να τις πούμε. Όπως σας είπα, υπάρχει μια έκθεση δραστηριοτήτων η οποία καλύπτει το διάστημα από τον Ιούνιο του 2008 μέχρι τον Μάιο του 2009. Αυτή είναι η τελευταία έκθεση που έχουμε υποβάλει. Όλα τα στοιχεία για το πότε κάναμε συνεδριάσεις, ποιους συναντήσαμε. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Βέβαια δεν θα επισέλθω σε αυτά αυτή τη στιγμή. Στην έκθεση αναφέρουμε και κάποια πράγματα για τα... Ε, καθήκοντά μας ως προς την ανεξαρτησία της Όλαφ και πώς μπορούμε να το παρακολουθούμε αυτό και γνωρίζουμε φυσικά και τι απειλές υπάρχουν για την ανεξαρτησία της Όλαφ κατά την ερευνητική της λειτουργία. Όπως σας είπα, ε, το πιο σημαντικό μας καθήκον είναι να διασφαλίσουμε ότι η Όλαφ κάνει τις έρευνά της με τον κατάλληλο τρόπο. Και αυτό φυσικά μας προδίδει τη βάση για να εκφράσουμε την άποψή μας για την ανεξαρτησία της Όλαφ ε, κατά την διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της. Αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε... Ε, αναφέρεται στην έκθεση. Πολύ μεγάλο τμήμα της έκθεσης είναι αφιερωμένο σε αυτό ακριβώς και έχουμε και κάποια στοιχεία για τις πληροφορίες και τα αρχεία που λαμβάνουμε από την Όλαφ πέραν των εκθέσεων που είναι υποχρεωμένοι να μας υποβάλει η Όλαφ. Ένα τομέα δραστηριοτήτων, τον οποίο θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό, είναι αυτέ οι εκθέσει των εννέα μηνών. Όπω σα είπα, η Όλαφ πρέπει να μας αναφέρει πότε και για ποιο λόγο μία ε, ε, έρευνα δεν κλείνει εντός των 9 μηνών. Το έχουμε ξανακάνει, έχουμε εκφράσει την άποψή μας για το 9 μηνό διάστημα. Θεωρούμε ότι το 80% όλων των υποθέσεων ε, συνήθως είναι άνω των 9 μηνών και τότε εξετάσαμε και για ποιο λόγο. Ε, οι υποθέσεις αυτές δεν ολοκληρώνονται ενός 9 μηνών και μετά εξετάζουμε. Αυτέ οι αιτιολογήσεις είναι σωστέ, είναι οι αυθεντικές αιτίε. Και ξέρουμε ότι περίπου στο μισό των περιπτώσεων όντω αυτό συμβαίνει, αλλά για τι υπόλοιπε, μάλλον δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αυτό το αναφέρουμε σαφώ στην έκθεσή μα. Λέμε ότι το τάδε δεν είναι σωστό, διότι οδηγεί σε λανθασμένα συμπεράσματα ω προ την αποτελεσματικότητα τη ε, έρευνα. Και ε, υπάρχουν φυσικά και πόροι ε, οι οποίοι μπορεί να έχουν δοθεί και μπορεί να είναι πολύ πιο δύσκολη η αξιολόγηση αν έχουμε κάποιες καθυστερήσεις ή όταν είναι τελείως στάσιμες οι έρευνες. Εξετάζουμε και κατά πόσον υπήρχε και επιρροή ε, στην Όλαφ. Προσπαθούμε να βρούμε ποια ήταν τα πραγματικά αίτια, για ποιο λόγο δεν ολοκληρώθηκαν εγκαίρως όλες αυτές τις υποθέσεις. Δεν υπάρχει βέβαια τίποτα τον οποίο να υποδεικνύει ότι οι καθυστερήσεις οφείλονται σε πίεση, ε, έλλειψη ανεξαρτησίας, αλλά μπορεί να υπάρχουν κάποιοι άλλοι παράγοντες οι οποίοι είναι υπεύθυνοι. Έχουμε λοιπόν εκθέσεις τις οποίες μας επιβάλλει η Όλαφ, ε, κάναμε και ανταλλαγές απόψεων επ' αυτών. Δεν νομίζω ότι έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Νομίζω όμως ότι έχω καλύψει το πιο σημαντικό τμήμα των εργασιών που πρέπει να διεξάγουμε εμείς. Ε, ε, ο έλεγχος και οι εκθέσεις είναι από τα πιο σημαντικά μας καθήκοντα. Φυσικά έχουμε και την προσωπική μας άποψη για το εγχειρίδιο ερευνητικών λειτουργιών της όλα αυτό έχουμε συζητήσει, κάνουμε τακτικές συζητήσεις επί του θέματος. Αυτό το εγχειρίδιο είναι κάτι το οποίο βελτιώνεται συνεχώς και φυσικά κανένας δεν είναι πάντα ικανοποιημένος, γι' αυτό προσπαθούμε ε, συνεχώς να το βελτιώνουμε. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες συστάσεις, τις οποίες ε, έχουμε στο τέλος της έκθεσης δραστηριοτήτων. Ε, οι συνάδελφοι θα αναφέρουν κάποια από αυτά. Ε, αν μου επιτρέπετε θα δώσω το λόγο στη Ρόσλιν Ράιτ που θα σας ε, δώσει και κάποια στοιχεία για κάποιες άλλες από τις δραστηριότητές μας. Κύριε Πρόεδρε, εξωτιμοί κύριε Βουλευτέ, ευχαριστώ για την ευκαιρία να σας μιλήσω. Σε δύο θέματα θα αναφερθώ. ήμουν εισηγήτρια για δύο θέματα της αιτήσεως έκθεσης. Το ένα είναι ο κανόνας de και πώς συμμορφώνεται με αυτό η Όλαφ. Και το λέει στρατηγικός σχεδιασμός των ε, ερευνών για τον Τεμίνιμις. Η Όλαφ δεν έπαιζε ανοχής μηδέν όσον αφορά τις οικονομικές παρατυπίες και εγκλήματα. Και έτσι είναι το σωστό. Το ότι υπάρχει πολιτική μηδενικής ανοχής δεν σημαίνει ότι η ολαφ και το λεει στρατηγικος σχεδιασμος των ερευνων για τον τεμινιμις η ολαφ δεν ανοχης μηδεν οσον αφορα τις οικονομικες παρατυπιες και εγκληματα και ετσι ειναι το σωστο το οτι υπαρχει πολιτικη μηδενικης ανοχης δεν σημαινει οτι η ολαφ πρέπει να μελετήσει την κάθε περίπτωση αν υπάρχουν άλλοι φορείς ή όργανα που θα ήθελαν να αναλάβουν την υπόθεση αυτή. Οι εσωτερικές έρευνες, η IDOC, είναι ένα τέτοιο όργανο που μπορεί και θέλει να αναλάβει ορισμένες τέτοιες περιπτώσεις που είναι λιγότερο σοβαρές κάτω από το κατόφλι. υποθέσεις συντεμήνες για μικρά χρηματικά ποσά. Στο εγκόλπιό τη και στις διαδικασίες η Όλεφ έχει το ένα κατόφλι της σοβαρότητας, της βαρύτητας για ποιες περιπτώσεις θα αναλάβει. Βέβαια η βαρύτητα δεν ορίζεται πουθενά. Είναι θέμα λοιπόν διακριτικής, διακριτικού ορισμού. Τι εμπίπτει στην κατηγορία του σοβαρού ή της βαρύτητας ή όχι. Σε 45 περιπτώσεις μελετήσαμε στη συγκεκριμένη περίπτωση διάρκεια της έκθεσης. Φυσικά όλες αυτές έχουν κλείσει οι υποθέσεις. Να δούμε πώς εφαρμόστηκε ο ορισμός της σοβαρότητας και επικύλει Ιδιαίτερα όσον αφορά εσωτερικές υποθέσεις. Η όλα ανταποκρίθηκε. Εμείς το βάλαμε στη γνωμοδότησή μας είχαμε θετική απάντηση από την Όλαφ. Πήραν πολύ στα σοβαρά τις ανησυχίες μας και θέλουν να εφαρμόσουν τις συστάσεις μας. Το συζητάμε τον κύριο Μανιέ που είναι επικεφαλής της IDOC. Οι αυτές του Γενικού Διευθυντή της Όλαφ και τον κύριο Μανιέ ήταν πάρα πολύ γόνιμες. Στο μέλλον, άλλες μικρές υποθέσεις που στο παρελθόν τις χειρίστηκε η Όλαφ, μπορεί να τις χειριστεί η IDOC. Τώρα, για εξωτερικές περιπτώσεις, πιο δύσκολο. Μερικές φορές δεν υπάρχουν όργανα που θα μπορούσαν να τις αναλάβουν. Και μόνο η Όλαφ μπορεί να ασχοληθεί με αυτές. Πιο δύσκολο αυτό για τις εξωτερικές περιπτώσεις. Το συζήτησα όμως με επικεφαλή των μονάδων στη Γενική Διεύθυνση Α και Β. Το γνωρίζουν το πρόβλημα και ακολουθούν επικοδομητική πρακτική, δηλαδή και οι πόροι δεν είναι πολλοί. Κατά την άποψή μας και την άποψη της Όλεφ θα πρέπει να επικεντρώνω την προσοχή πιο σοβαρές περιπτώσεις όπου το έχουν κίνδυνο τα οικονομικά της Ένωσης και μη στρέφουν πόρους προς περιοχές που μπορούν να, αναλάβουν, να τις αναλάβουν άλλοι. Συμφωνούμε σε αυτό. Αυτά για τα ντεμίνιμες. Το δεύτερο είναι ο στρατηγικός προγραμματισμός των ερευνών. Αυτό συνεχίζεται. Είναι σε εξέλιξη. Δεν έχουμε γνωμοδοτήσει για την ώρα, αλλά το έχουμε συζητήσει με τους επικεφαλείς μονάδων και στο διοικητικό σκέλος Α και Β της Όλαφ πώς σχεδιάζουν τις υποθέσεις τους, πώς χρησιμοποιούν τους ανθρώπινους πόρους. Η ΟΛΑΦ προγραμματίζει οι έρευνες και να έχουν την καλύτερη χρήση των λιγοστών πόρων εξάλλου που έχουν. Εντυπωσιάστηκα από το πώς σχεδιάστηκαν πολλές έρευνες. Αυτό είναι μια δουλειά που συνεχίζεται. Στους επόμενους μήνες θα κάνουμε μια γνωμοδότηση προς την Όλαφ. Το πνεύμα συνεργασίας μεταξύ μας είναι πάρα πάρα πολύ καλό. Θέλουν τη βοήθειά μας. του χρόνου πιστεύω να μπορώ να σας μιλήσω πάλι με το ίδιο θετικό πνεύμα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ε, ο πρόεδρος της, ε, της εποπτείας παρακαλεί τον κύριο Γιώργη, να δοθεί ο λόγος στον κύριο Γιώργη να πει και αυτός κάτι. κύριε Πρόεδρε. Η αρμόδιότητά μου είναι για περιπτώσεις που αφορούν τις ε, εθνικές αρχές δικαιοσύνης, που διαβάστηκαν δηλαδή προς τις εθνικές αρχές. Είναι γνωστό ότι η Όλαφ δεν είναι δικαστικό όργανο, Η Όλαφ δεν μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις. Μπορεί όμως να βοηθήσει οι εθνικές αρχές να το κάνουν αυτό. Στην έκθεση έχουμε, όπως βλέπετε, ελέγχθησαν 36 εκθέσεις έρευνας που εστάγησαν μέσω της Όλαφ στις ε, εθνικές δικαστικές αρχές. Αυτές οι εκθέσεις έρχονται στο τραπέζι των συνεδριάσεων της ε, Επιτροπής Υποπτίας και δίνονται και στην Όλαφ. Η Επιτροπή Εποπτείας κάνει μια πρώτη ανάλυση αυτών των ε, εκθέσεων και συζητάει το περιεχόμενό της με τον ΟΛΑΦ να δούμε κατά πόσο είναι σκόπιμο να γίνει αυτή η έρευνα Η Επιτροπή Εποπτείας ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την ποιότητα της έκθεσης και περιπτώσεις που δεν θα ακολουθηθούν, παρακολουθηθούν μάλλον από τις εθνικές αρχές. Γι' αυτό ερευνήσαμε πολλές περιπτώσεις του παρελθόν. όπου υπήρχε κίνδυνος παραγραφής. Επίσης, στις εκθέσεις Ε, Λίγες ήταν οι εκθέσει όπου υπήρχε ο κίνδυνος παραγραφής λογοδράση των εθνικών αρχών. Περισσότερο, το πιο ενδιαφέρον είναι να βελτιωθεί η ποιότητα των πληροφοριών των εκθέσεων μέσω της ανάλυσης των υποτιθέμενων ε, καταδικαστέων περιπτώσεων. Σε πολλές περιπτώσεις οι εκθέσεις έρευνας ελέγχθησαν από την Επιτροπή Εποπτείας αφού προηγουμένως είχαν ήδη είχε σταλεί ο φάκελος στις Εθνικές Δικαστικές Αρχές. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε ήδη αποφασίσει ότι αυτά είναι παράβαση. του κανονισμού 1037 του 99 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναφέρει ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων των ενδιαφερομένων πείτε αν τα έγραφα αυτά διαβαστούν πολύ νωρίς. Καταρχήν όμως η Επιτροπή Εποπτείας πρέπει να μείνει μέσα στα πλαίσια της εντολής με βάση το 1063 όπως σας είπα. Αυτό αναφέρεται ιδιαίτερα στη νομική υποχρέωση της Επιτροπής Εποπτείας. Δεν, αφορά τις, ε, δεν πρέπει εμείς να δράσουμε στη διάρκεια των ερευνών της ΟΛΑΦ ούτε να λάβουμε δράση αυτόνομα για θέματα που αφορούν εκθέσεις που έχει στείλει η Όλαφ στις εθνικές δικαστικές αρχές και ακόμη κρεμούν. Πρέπει να μελετάμε κάθε περίπτωση τι πρέπει να γίνει. Φυσικά η γραμματεία ήδη επιβαρύνεται από τον φόρτο εργασίας. Δεχομένως λοιπόν να ασκήσουμε έφεση κατά του, της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Εν πάση πτώση, προκειμένου να αμφισβητήσουμε την απόφαση του δικαστηριού, θα πρέπει να εισαχθούν νέες μέθοδες συνεργασίας με την Όλαφ διότι θέλουμε να προστατευτούν τα θεμελιώδη δικαιώματα στη διάρκεια της έρευνας. Αυτό είναι η υποχρέωση της ε, Επιτροπής Εποπτείας. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι αναδρομικά να ερευνήσουμε κατά πόσον σημειώθηκε παράβαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και οποιοδήποτε σχόλιο όμως στην περίπτωση αυτή δεν θα έχει πρακτική σημασία. Πέντε εργάσιμες μέρες απαιτούνται προκειμένου να μεταφερθεί το, να σταλεί το υλικό από την Όλαφ στις εθνικές αρχές. Η Επιτροπή Εποπτείας προτείνει η Όλαφ να ζητάει απόφαση για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση προκειμένου να δούμε, να δει αν τηρήθηκαν τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι διαδικασίες, οι εγγύησεις όσον αφορά τις διαδικασίες. Σε περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες και επιφυλάξεις, Ε, τότε έχει ε, πρόσβαση σε ε, όλο το φάκελο της ανάκρισης και της έρευνας. Η Επιτροπή μας θέλει πάντα να βεβαιώνεται ότι λαμβάνονται υπόψη τα παράπονα και οι καταγγελίες των ενδιαφερομένων για παραβίαση δεδομένων και προσωπικών δικαιωμάτων. Ε, ε, τις διαδικασίες ε, που έχει ελέγξει, στοιχεία που έχει λάβει η Όλαφ. Και εδώ εννοεί η Επιτροπή Εποπτείας όλες τις περιπτώσεις, όχι μόνο αυτές που εκκριμούν στην εθνική δικαιοσύνη του κάθε κράτους, ακόμα και σε περίπτωση υποτιθέμενης, εικαζόμενης παραβίασης δικαιωμάτων. Και γι' αυτό και ο διαμεσολαβητής ε, και οι άλλες αρμόδιες αρχές έχουν επιμείνει πάρα πολύ ότι θα πρέπει ο Όλαφ να ε, προσέχει και να τηρεί αυστηρά τους κανόνες. Αυτά λοιπόν για την έκθεση δραστηριοτήτων και το τομέα ε, αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Εποπτείας της Όλαφ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ωραία, ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο στον εισηγητή, στην εισηγήτρια, συγγνώμη, κυρία Γκρέσλε. Ευχαριστώ πολύ την κυρία και τους κυρίους ε, της Επιτροπής Εποπτείας για την ενδιαφέρουσα και σημαντική αυτή έκθεση. Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε σε ένα ενδιαφέρον σημείο για τα διορθωτικά ταμεία ε, Ακούσαμε τα διαρθωτικά ταμεία, ακούσαμε την εξωτερική βοήθεια και τώρα φτάσαμε στο τρίτο, λέω, ενδιαφέρον θέμα για την καταπολέμηση της απάτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση της Επιτροπής Εποπτείας κατέδειξε και σε εμά ότι υπάρχουν προβλήματα, ότι εργάζονται ε, και λειτουργεί το οικοδόμημα ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μπορεί να μην λειτουργεί άψογα, λειτουργεί όμως. Και εκεί όμως που σταματάει να λειτουργεί είναι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να μπουν στο παιχνίδι τα κράτη-μέλη. Το τελευταίο διάστημα ασχοληθήκαμε πολύ εντατικά με το θέμα του κανονισμού 1073 ε, του 99. Έχουμε και 11 παρακαλώ έγγραφα εργασίας έκτοτε. Ε, μας τα παρουσίασε και η Επιτροπή Εποπτείας και αν θέλει κάποιος νέος συνάδελφος να τα διαβάσει μπορεί να τα βρει στην ιστοσελίδα της Κοκομπού. Αλλιώς ελάτε στο γραφείο μου. Και θα πρέπει να ασχοληθούμε με το εξή ερώτημα. Τι γίνεται με την καταπολέμηση της απάτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πού το πάει. Τώρα έχουμε οδηγηθεί σε αποτελμάτωση. Πέρσι το Νοέμβριο εγκρίθηκε η έκθεση και έκτοτε μηδέν ιστοπηλίκων. Η ε, ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρόλο που η Τσεχική Προεδρία ήθελε να δώσει συνέχεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κάνει τίποτα. Πού βρίσκονται τα προβλήματα, να σας πω. Μόλις 7% των περιπτώσεων που εξετάζει η Όλαφ και διαβιβάζει ε, στη δικαιοσύνη των κρατών επτών, μόλις το 7% καταλήγουν σε δικαστική απόφαση. 7%! Δηλαδή το 93% των περιπτώσεων της Όλαφ που εμείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τόσο προσοχή ε, χειριζόμαστε και προσπαθούμε να τηρούμε και τα δικαιώματα και τα πάντα, ε, είναι άσκοπα γιατί ε, τα κράτη-μέλη ε, ολιγορούν και προστατεύουμε τελικά εγκληματίες. Φέτος το Φλεβάρι υπάρχει ένα έγγραφο εργασίας δικό μου που συζητήσαμε εδώ. Έχουμε τα πρώτα στατιστικά στοιχεία ε, που μας έδωσε η Όλαφ για το θέμα αυτό. Και τι δείχνει η έκθεση. Ότι υπήρξαν και πολύ λίγες αθωώσεις στο 7% των δικαστικών αποφάσεων. Δηλαδή πραγματικά η Όλαφ ασχολείται με θέματα που πρέπει να ε, επιληφθεί δικαιοσύνη και αν θέλουμε ε, πραγματικά να σταματήσουμε κάποιους παρανομούντες ε, πρέπει να αναρωτηθούμε ποιο είναι ο αποδέκτης των παραπώνων. Το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο μέχρι τώρα δεν έχει καμία δομή για την καταπολέμηση της απάτης. Στη δική μου έκθεση που ξέρουν οι παλιοί συνάδελφοι ότι η Ονομέλεια πέρασε με 95%. Ε, υποχρεώνουμε το Συμβούλιο να κάνει δομές για τη συνεργασία μαζί μας και με την Όλαφ και να θεματοποιήσει αυτό το ζήτημα της ε, καταπολέμησης της απάτης, δηλαδή να ασχοληθεί με αυτό. Τίποτα το Συμβούλιο, όπως και το 93% των περιπτώσεων τη Όλαφ που δεν δίνεται συνέχεια. Γι' αυτό ε, θέλω να σας πω ότι και η σημερινή συζήτηση με την Επιτροπή Εποπτείας θα πρέπει να είναι αφορμή και για μας να ε, ε, στείλουμε τις ευθύνες εκεί και να αποδώσουμε τις ευθύνες εκεί που ανήκουν, δηλαδή στα κράτη-μέλη. Να δίνουν συνέχεια στις περιπτώσεις της Όλαφ. Και στη Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει θα τη βάλουν στα τελωνία, τέρμα Θεού. μια απόφυση θα είναι στην Επιτροπή η υπηρεσία αυτή. Ο Επίτροπος μου είναι προσωπικά πάρα πολύ συμπαθής, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορεί να συνεργαστεί η Όλαφ. Και δεν είναι και πλέον αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα πρέπει κάποιος να μου εξηγήσει τι έγινε. Πριν από 10 χρόνια, μετά από πίεση του Κοινοβουλίου, ιδρύθηκε η Όλαφ. Αν δεν προσέξουμε τώρα, και υλοποιήσει ο πρόεδρος τα σχέδιά του, δηλαδή την πετάξει έξω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αν δραστηριοποιείται μόνο εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή της το ζητήσει να το κάνει, ε, τότε να ξεχάσουμε τις εσωτερικές έρευνες, να ξεχάσουμε έρευνες που αφορούν την ίδια την Επιτροπή και να ξεχάσουμε ακόμα περισσότερο τη συνεργασία με τα κράτη-μέλη, γιατί ως Κοινοβούλιο δεν θα έχουμε κανένα μέσο πίεσης πλέον. Τα παρακαλούσα λοιπόν τους ε, κυρίους και τις κυρίες ε, της Επιτροπής Εποπτείας να μας πούν πώς το βλέπουν. Τι είναι αυτή η εξωτερήκευση της Όλαφ, γιατί την, την εξαιρούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το έχετε συζητήσει, θα το συζητήσετε, διότι στο θέμα αυτό θα πρέπει να είμαστε όλοι ε, στοιχημένοι, συμπαγείς, να δούμε πώς θα λύσουμε τα προβλήματα. Το θέμα της μακροχρόνιας διαδικασίας 9 μήνες και πλέον στο 75% των περιπτώσεων, συν την απροθυμία των κρατών μελών για συνεργασία, είναι πρόβλημα. Έχουμε πολλά προβλήματα γιατί αρνείται τη συνεργασία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παραμένει το πρόβλημα της μη πρόσβασης ε, στη βάση των δεδομένων από την Όλαφ όπου κάθε φορά γίνονται εκτενείς ερωτήσεις και αιτήσει και χρονοβόρες και σε τελική ανάλυση τα προβλήματα παραμένουν και τα βρίσκουμε μπροστά μας. Η Επιτροπή Εποπτείας το ανέφερε τα τελευταία δύο-τρία χρόνια είχαμε αποφάσεις ε, του πρωτοδικείου στο Λουξεμβούργο και η πιο πρόσφατη ήταν ολέθρια. Διότι δημιουργεί δύο κατηγορίες ανθρώπων. Τους κοινοτικούς υπαλλήλους και τους υπολείπους θνητούς. Γιατί γίνεται λόγος για καλύτερη αντιμετώπιση των κοινοτικών υπαλλήλων σε σχέση με του υπόλοιπου θνητού. Και όταν σε έχουν εκλέξει υπόλοιποι θνητοί, δεν μπορεί να το δέχεσαι αυτό. Αλλά αν δεν μπορεί να αλλάξει ούτε τη νομική βάση, ε, είναι τα χέρια σου δεμένα. Και δεν έχουμε την ευκαιρία. Και μάλιστα είχε τεθεί και ζήτημα να κάνει έφεση η Όλαφ για αυτό το ζήτημα. Άντε να το εξηγήσει αυτό στους ψηφοφόρους σου μετά. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν φυσιολογικοί άνθρωποι και να έχουν ε, αντιμετώπιση κοινών θνητών και μετά υπάρχουν κάποιοι που ε, απολαμβάνουν πολύ ε, περισσότερων προνομίων που είναι κοινοτικοί πάλι. Βλέπουμε με ικανοποίηση ότι η Επιτροπή Εποπτείας κάνει καλά τη δουλειά της. Ανισχώ γιατί από ό,τι φαίνεται το εγχειρίδιο της Όλαφ ακόμα να τελειώσει. Γιατί, τι είναι αυτό το εγχειρίδιο. Δεν μπορούμε να το κλείσουμε αυτό το εργοτάξιο. Στην Επιτροπή Εποπτείας ξέρουμε ποια είναι τα προβλήματα που πρέπει να λυθούν. Η διαβίβαση των ε, εγγράφων, ας πούμε, στη δικαιοσύνη των κρατών μελών. Η Επιτροπή Εποπτείας συνεργάζεται και πρέπει να συνεργαστεί με την Όλαφ για να λυθεί το θέμα. Εμείς από το Κοινοβούλιο δεν μπορούμε να το λύσουμε, ούτε είναι ο ρόλος μας και η δουλειά μας. Αν ε, όμως θέλετε να αφήσουμε την Όλαφ να λειτουργήσει καλά και να δουλέψει και το Συμβούλιο Εποπτής. Πρέπει να τους αφήσουμε να συνεργαστούν. Δεν έχω καταλάβει ότι υπάρχουν μεγάλα προβλήματα ούτε από όσα άκουσα ούτε από όσα διάβασα. Έχουν καλή συνεννόηση. Αν δεν έχουν να μα το πούν, αν δεν μπορούν να βρουν μεταξύ τους δηλαδή μια λύση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χατζημαρκάκη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω για την έκθεση αρμοδιοτήτων και που μας παρουσίασαν και προφορικά. Είναι καλή έκθεση, καλά διαρθρωμένη, καλά τα κεφάλαια και μπορούμε πολύ να κατατοπιστούμε. Εσείς είστε σημαντικοί για τη διαφύλαξη της ανεξαρτησίας της Όλαφ. Γι' αυτό ε, ο τρόπος με τον οποίο συνεργάζεστε με την Όλαφ αλλά και με εμά είναι αποφασιστική σημασίας. Αλλά ίσως και πέρα αυτό που είπε η κυρία ε, Γκρέσλε, εγώ θεωρώ ότι όσο πιο ανεξάρτητη από την Κομισιόν είναι η Όλαφ, τόσο το καλύτερο. Εμένα δεν με νοιάζει αν είναι παρά το αντιπροέδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή όχι η Όλαφ. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι ανεξάρτητη. Όσο πιο ανεξάρτητη είναι, τόσο πιο αξιοσέβαστη είναι και τόσο καλύτερα είναι. Και παίζετε εσεί εκεί η Επιτροπή Εποπτεία ρόλο. Σε μεγάλο βαθμό εγώ θέλω να επενέσω και το έργο της Όλαφ και, και χαίρομαι γι' αυτό για μας ως εμπνευστέ ή εφευρέτε τη Όλαφ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ωστόσο, υπάρχουν δύο ενότητε προβληματικέ. Πρώτον, η παραγραφή διαφόρων περιπτώσεων υποθέσεων στη δικαιοσύνη. Όταν ε, ερευνούν και διώκουν ε, τα κράτη-μέλη έχουμε λιγορίες και χρονοτιβές και παραγράφονται τα αδικήματα. Και όπως είπε η κυρία Γκρέσλε, είπε 7% μόλις, όχι 9, 7% έχουμε δικαστική απόφαση. Ε, είναι ολέθριο αυτό. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Ότι πολλές φορές είναι εικονικό φάρμακο η Όλαφ για τα μάτια. Και υπάρχει εννιάμινη, λέει, προθεσμία που είναι τόσο σημαντική για τη δουλειά σας και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να την υπερβαίνουμε. Και διαβάζω στην έκθεσή σας όμως ότι σε 80 περίπου των περιπτώσεων, τις 100 των περιπτώσεων, υπερβαίνουμε αυτή τη διαδικασία. Μα αν μια διαδικασία διαρκεί πάνω από 9 μήνες θα πρέπει να σας ενημερώνουν. Ερωτώ, σας ενημερώνουν όντω πάντα γιατί από την έκθεση αντιλαμβάνομαι ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο και είναι πάρα πολύ αμφίβολο αυτό γιατί αυτή είναι η αρχή του τέλους, η αρχή της παραγραφής και της κατρακύλας και δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό. Τι μπορείτε λοιπόν να κάνετε πολύ συγκεκριμένα στη δουλειά σας, στη συνεργασία με την Όλαφ για να τηρείτε το ένα άμυνο. Το δεύτερο σύνολο των προβλημάτων αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα και αυτό είναι βασική σας αποστολή. Τα θεμελιώδη δικαιώματα των υπόπτων κατά τη διάρκεια της ε, ε, Διαδικασία να γίνονται σεβαστά. Αυτά όμω είναι ανδρομικά γιατί εσεί δεν μπορείτε κατά τη διάρκεια τη διαδικασία όταν κρεμεί τη δικαιοσύνη να επεμβαίνετε. Ο κύριο Γεώργη μα εξήγησε ε, εκτενώς ότι θα αλλάξει και πρέπει να αλλάξει η διαδικασία αυτή. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει πρώτερη ενημέρωση ακόμα και δεν επιτρέπεται να έχετε πρόσβαση στις ε, υποθέσεις, τουλάχιστον να τις γνωρίζετε. Αλλιώς πώς θα διαφυλάσσονται τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και ως πολιτικοί εμείς γνωρίζουμε ότι άμα σε κατηγορήσουν για κάτι μία φορά, και σήμερα στο διαδίκτυο αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο, σου μένει ρετσινιά. Και σε καταδικάζουν από χέρι, ακόμα και αν δεν έχεις κάνει τίποτα. Τώρα είμαστε δηλαδή σε πάρα πολύ ολιστηρό έδαφος. Γι' αυτό, συγκεκριμένη ερώτηση. Ενημερώνεστε για όλες τις περιπτώσεις που έχουμε παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων οι επεμβάσεις ή απλώς σε περιπτώσεις και υποθέσεις που διαβιβάζονται ε, στα κράτη-μέλη και στα εθνικά δικαστήρια. Ευχαριστώ πολύ. Euh, ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα η έκθεση. Και ελπίζω στη συζήτηση να ξεχωρίσουμε τα σφάλματα και τις απάτες τη συζήτηση που είχαμε το ελεκτικό συνέδριο. Δεν είναι δουλειά του ελεκτικού να αναζητήσει συστηματικά τι απάτες, διότι δηλαδή, οι απάτες τεχνικά δεν είναι το άθροισμα των λαθών. Και μέσω των σφαλμάτων δεν καταλήγει κανείς κατά ανάγκη πάντα στην απάτη. Σημαντική αυτή η διάκριση. Με διέφερε ιδιαίτερα το τελευταίο πόρισμα ε, συμπέρασμα για το συγκεκριμένο ποσοστό. Τι να πω, οι έρευνες της Όλαφ δεν έγιναν σωστά, δεν καταλήγουν κάπου ή υπάρχει πρόβλημα των εθνικών δικαστικών αρχών. Και μετά τα μέσα που διαθέτει η υπαρχει προβλημα των εθνικων δικαστικων αρχων και μετα τα μεσα που διαθετει η Στην έκθεσή σας λέτε όχι πλέον προσωπικό. Γιατί όχι. Εμείς στο Ευρωκοινοβούλιο, αρχή του προπολογισμού, αν κρίνουμε ότι χρειάζονται επιπλέον πόροι στο ελεγκτικό, στην Όλαφ για τις όλες τις ερωτήσεις προς τους Επιτρόπους. Η πρώτη ερώτησή μου είναι έχετε απάτη, απάτες και γενικά όλοι απάντησαν όχι πολλέ. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι υπάρχουν απάτες, περισσότερες από ό,τι φανταζόμαστε, διότι ο απαταιώνας δεν κάνει σφάλματα. Έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα λοιπόν στην απάτη και αν αύριο απαιτήσετε επιπλέον πόρου, φέρτε μας τι αποδείξεις και θα βρεθεί η πολιτική πλειοψηφία να υπάρξουν τα επιπλέον μέσα. Μετά τα 500 πρόσωπα προσωπικό της Όλαφ, 180 είναι στη γραμματεία και στις γενικές υποθέσεις και 170 άτομα στις έρευνας. Δεν ξέρω πώς διαχειρίζεται την έρευνα. Αν 180 στη γραμματεία και 170 στην έρευνα, είναι σωστή αυτή η κατανομή των ανθρώπινων πόρων όσον αφορά την έρευνα ή μήπως θα πρέπει να βάλετε περισσότερα άτομα στην έρευνα και λιγότερο στα γραφεία. Και επανέρχομαι στην προηγούμενη ερώτηση. Σε επαρκούν οι ανθρώπινοι πόροι που διαθέτεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα από τα βασικά συμπεράσματα της Επιτροπής Εποπτείας είναι ότι υπάρχουν άμεσες και έμεσες απειλές για την ανεξαρτησία της Όλαφ στη διεξαγωγή των ερευνών. Αυτό είναι συμπέρασμα αρκετά οξύ, άμεσες και έμεσες και, και υπόγειες ενδεχομένω. Ως πρώτο συμπέρασμα ε, αξίζει τον κόπο να ασχοληθούμε περισσότερο με αυτό. Στην έκθεσή σας αναφέρετε και μερικά παραδείγματα για το πώς αυτές οι απειλές ε, υλοποιούνται και σάρκα και οστά. Και πώς μπορεί κανείς να αντισταθεί σε αυτές τις ε, απειλές αν προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κάτι που σας έχει απασχολήσει. Τι κάνετε, εσείς κάνετε έκθεση μετά. Έχετε πειθαρχικές διαδικασίες ή και δικαστικές. Έχετε συγκεκριμένα παραδείγματα. Όταν διαπιστώνετε τέτοιες απειλές κατά της όλαφα από πλευρά θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μια ερώτηση που την κάνουν κάποιε φορές συνάδελφε για τι έρευνε της Όλαφ. Η κυρία Γκρέσλε είπε ότι φαίνεται να υπάρχει έλλειψη συνεργασία με τις εθνικέ δικαστικές αρχές ή δεν υπάρχει επαρκής ε, διοικητική ικανότητα, πούμε, όπως ανάφερε ο κ. Σουγγί. ποιο είναι ο λόγο, για τον οποίο έχουμε τόσες πολλές περιπτώσεις που έχουν πολύ μακρά περίοδο έρευνας. Πρόεδρος, έχω και εγώ μερικές ερωτήσεις. Και επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα παρακαλέσω τον πρόεδρο να απαντήσει με γητό τρόπο, αλλά μπορείτε να μας απαντήσετε στα υπόλοιπα γραπτά. Συμφωνώ με τον αντιπρόεδρο Ντίβ η εμπειρία μας δείχνει ότι οι καλύτεροι απατεώνες σέβονται τους τύπους. Όταν τηρείται ο τύπος δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν απάτες. Είχαμε και διμερή αλλαγή απόψε με τον Πρόεδρο. Σήμερα θέτω ορισμένα ερωτήματα στην Επιτροπή μας. Μπορείτε να μας πείτε τι δεν πάει καλά στην Όλαφ που υπάρχουν σκιές ή ποιο είναι το επίπεδο διαφάνειας στην Όλαφ. Ο συνάδελφος Χατζημαρκάκης πριν μας μίλησε για το επίπεδο ανεξαρτησίας. Υπάρχει πραγματική ανεξαρτησία μεταξύ Όλαφ και Επιτροπής ή μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση. Τι λύσεις υπάρχουν και επίπεδο ανεξαρτησίας όχι μόνο ως προς την Κομισιόν, ως προς τα άλλα όργανα της Ένωσης και ανεξαρτησίως προς τα κράτη-μέλη. Άλλη ερώτηση. Ελέγξατε τις διαφορές στη μεταχείριση της Όλαφ από τα 27 κράτη της Ένωσης. Υπάρχει ομοιομορφία της δράσης της Όλαφ έναντι όλων των κρατών. Κάτι άλλο λεπτό θέμα. Τι βαθμό συνεργασίας υπάρχει μεταξύ της Όλαφ και των δικαστικών πιο συγκεκριμένα εθνικών αρχών και αν μπορεί να γίνει κάτι γι' αυτό. Σε αυτό συμφωνώ με αυτό που είπε πριν η Στέφος Γκρέσλε για την Κομισιόν πρέπει να ασκηθεί πίεση στο Συμβούλιο και την Κομισιόν να παρεμβαίνουν ως προς τα εθνικά κράτη που δεν εγγυώνται επαρκή συνεργασία με την Όλαφ για να πετύχουν ένα καλό αποτέλεσμα έρευνας για τις απάτες. Πολλοί συνάδελφοι κάναμε πολλές σημαντικές ερωτήσεις. Σας δίνω το λόγο κύριε Πρόεδρε. Έχουμε άλλη μία, συνεχίζει η συνεδρίασή μας και θα περιμένουμε το συμπλήρωμα των απαντήσεών σας γραπτά για καλύτερη συνεργασία στο μέλλον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και όλα τα υπόλοιπα μέλη που έθεσαν ερωτήσεις και μας έκαναν παρατηρήσεις και σχόλια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας να έχουμε τα στοιχεία αυτά. Θα απαντήσω λοιπόν κάποιες από τις ερωτήσεις. Είναι στενά τα χρονοδιαγράμματα, οπότε θα απαντήσω πολύ επιφανειακά. Ξέρετε ότι η Όλαφ ε, είναι εκτός Ευρωπαϊκής Επιτροπής και βρίσκεται απ' έξω. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο συζητάτε από εμά ε, αυτή τη στιγμή. Πρόκειται για μια νέα πρόταση. Προφανώς θα τη συζητήσουμε αυτές τις προτάσεις ε, πολύ στενά. Δεν έχουμε άποψη επί του θέματος για τα υπέρ και τα κατά. σαφώς θα το παρακολουθήσετε ένα Επιτροπή Εποπτείας διότι ε, αφορά και εμάς και το ρόλο της Όλαφ και τις δραστηριότητες πολέμηση από αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό τους. Όσον αφορά τώρα στην πρόσβαση, υπήρξε κάποια σχετική ερώτηση για την πρόσβαση που έχουμε σε πληροφορίες, έγγραφα, συστήματα υπολογιστών κλπ. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι μέχρι τώρα πάντα μας έδιναν αυτό που ζητήσαμε και φαντάζομαι ότι και στο μέλλον πάντα θα λαμβάνουμε αυτά που ζητάμε. Ορισμένες φορές μπορεί να καθυστερήσει λίγο, αλλά συνήθως λαμβάνουμε τις πληροφορίες που ζητούμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα. Τώρα, ερώτηση για το κατά πόσο είναι ανοιχτή σε πληροφορίες, ε, κατά πόσο μαθαίνουμε ε, τι γίνεται με τις υποθέσεις που είναι άνω των 9 μηνών. Ε, ναι, αυτό πιστεύουμε. Αν δεν έχουμε λάβει πληροφορίες, συνήθως είναι διοικητικό λάθος. Ε, πάντα ε, τις βρίσκουμε όμως αυτές τις υποθέσεις οι οποίες κρατούν πάνω από 9 μήνες. Αν μαθαίνουμε για όλες τις υποθέσεις, στις οποίες έχει υπάρξει παραβίαση θεμελιωδών και διαδικαστικών δικαιωμάτων. Εδώ δεν μπορώ μάλλον να σας απαντήσω θετικά. Ορισμένε φορές λαμβάνουμε και την απόφαση από το δικαστήριο ε, αλλά και η Όλαφ έχει δικές της εσωτερικές δομές για να ασχολείται με τα θέματα αυτά. Το σκεπτικό είναι να προσπαθήσουμε να έχουμε στοιχεία από όλα αυτά. Η κυρία Γκρέσλε αναφέρθηκε και στις έρευνες οι οποίες οδηγούν σε ένα πολύ μικρό ποσοστό δικαστικών αποφάσεων στα κράτη-μέλη. Είναι πολύ δύσκολο να εξετάσουμε στατιστικά στοιχεία υπό αυτή την έννοια. Δεν έχουμε εξετάσει προς το παρόν στατιστικά στοιχεία. Αυτό που πρέπει να εξετάζουμε εμείς είναι πώς διαβιβάζονται οι υποθέσεις ε, στα κράτη-μέλη και πώς παρακολουθείται η διαβίβαση αυτή. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να εξετάζουμε εμείς, να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί με αυτές τις υποθέσεις. Και ο βασικός ε, ρόλος μας είναι να δούμε αν καθυστέρησαν με τον ένα με τον άλλο τρόπο αυτές οι υποθέσεις. Ο κίνδυνος όμως ε, έχει μειωθεί. Το έχουμε εξετάσει και η απάντησή μας σε αυτό είναι σαφής. Ως προς τους κινδύνους για την Όλαφ, συγκεκριμένους κινδύνους, αυτό που λέμε στο συμπέρασμα 1 του εγγράφου είναι ότι Εντοπίζουμε δυνητικές ε, πηγές απειλής, ε, δεν μπορούμε να βρούμε τι δυνατότητα έχουν ε, να βλάψουν την ανεξαρτησία της Όλαφ. Ο τρόπος με τον οποίο διεξάγουμε εμείς τη δουλειά μας είναι να γνωρίζουμε ότι μπορεί να υπάρξει ένα τέτοιο ενδεχόμενο και θα πρέπει να έχουμε μεθόδους να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία που διαθέτουμε και καταδεικνύουν ότι όντως συμβαίνει κάτι τέτοιο. Όσο για την ε, ε, ερώτηση που έθεσε ο πρόεδρος ε, στο τέλος, είναι τεράστιο το θέμα για το τι δουλεύει και τι δεν δουλεύει στην Όλαφ, αλλά κατά την άποψή μας σε γενικές γραμμές τα πράγματα δουλεύουν καλά. Δεν υπάρχει κάποια ενιαία προσέγγιση από πλευράς κρατών μελών για την Όλαφ, όλα είναι αναϋπόθεση. Όταν η Όλαφ ε, περνάει τις ε, έρευνές της ε, στις αρχές των κρατών μελών, εμείς κατανοούμε ότι τις αναλαμβάνουν και τις αντιμετωπίζουμε σοβαρότητα. Αυτή την εντύπωση έχουμε τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει κάτι. Χάθηκε το μικρόφωνο του ομιλητή. Ελπίζω να μην ξέχασα πολλά πράγματα και με συγχωρείτε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αν ε, μας δώσετε και κάτι γραπτός, διότι έγιναν και άλλες ερωτήσεις και φυσικά σας ζητήθηκαν και κάποια άλλα πράγματα και επειδή εμείς θεωρούμε πάρα πολύ σημαντική τη δουλειά σας, θα θέλαμε κάποια επιπλέον στοιχεία γραπτός. Να περάσουμε τώρα. Σας χαιρετώ σας, ε, σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Είστε επανειδήν. Να περάσουμε στο σημείο 8 της τη διάταξης. Πολύ σύντομα να πω λίγα πράγματα στους αδέλφους για τη συνεδρία των συντονιστών που έγινε χθε. Καταρχάς, ε, να ζητήσω ως πρόεδρος Επιτροπής της πολιτικές ομάδες να διαβιβάσουν στη γραμματεία τη θέση τους για ένα αίτημα για έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας για τις υπηρεσίες. Για το σημείο 2, το gender mainstreaming, το έχει αναλάβει ο αντιπρόεδρος ε, Στάες και εγώ θα αποστείλω μια επιστολή στον κύριο Σβένσον διαβιβάζοντάς του το όνομα του κυρίου Στάες στην κυρία Σβένσον. Επίσης, τι θα κάνουμε με τους ε, whistleblowers, τα επιστολές που φτάνουν στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού και παρουσιάζουν ε, συμπεριφορά που θα μπορούσε ίσως να ενδιαφέρει την Όλαφ. Ε, έχουμε καθορίσει μία διαδικασία μέσω της οποίας μπορούμε να κοινοποιούμε στην Όλαφ ε, όλες αυτές τις επιστολές και τα στοιχεία που φτάνουν στην Όλαφ. Αυτό είναι κάτι το οποίο είχαμε κάνει και στο παρελθόν. Οι πολιτικές ομάδες επίσης δεσμεύτηκαν να διαβάσουν στη Γραμματεία τα ονόματα των βουλευτών που θα συμμετάσχουν στις αντιπροσωπείες για το 2010 στην Ελλάδα, την Κροατία, την Ουγγαρία και στην Ιταλία. Είναι επίγον κυρίως ε, να μας πείτε ποιοι θα πάνε στην Ελλάδα. Ε, εγώ θα προεδρεύσω τις αποστολής στην Ελλάδα διότι υπάρχει μια σχετική συζήτηση και το ταξίδι θα γίνει στο τέλος Απριλίου. Ένα εξίσου σημαντικό θέμα το οποίο συζητήσαμε χθε είναι πώς πρέπει να κινηθούμε, τι στάση πρέπει να κρατήσει η Επιτροπή μας σε αυτή τη φάση που τίθεται σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας. Διότι όλοι λίγο πολύ και ο Πρόεδρος και οι συνάδελφοι συντονιστές διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μια γενική τάση να μείνει στο περιθώριο η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Γι' αυτό αποφασίσαμε ότι δεν μας αρέσει αυτό. Ε, παρουσιάσαμε και τα επιχειρήματά μας. Εγώ το έχω πει προφορικός και στον πρόεδρο Μπούζεκ σε μια συνάντηση που είχαμε και επισήμως ε, στην διάσκεψη των προέδρων των επιτροπών και αποφασίσαμε ότι θα αποστείλουμε μια επιστολή στον ε, πρόεδρο Μπούζεκ και στον πρόεδρο Λένελ για την ε, διαδικασία που απαιτεί ταχεία διαδικασία για τον ε, προϋπολογισμό και η, ο ρόλος, το ρόλο της Επιτροπής του Ελέγχου του Προϋπολογισμού μετά τη θέση της Συνθήκης της Λισαβόνας. Ξέρετε ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας αναγνωρίζει το νομοθετικό έργο ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ένα από τα πιο σημαντικά είναι η Επιτροπή Προϋπολογισμός και η, Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Θεωρούμε λοιπόν ότι οι αρμοδιότητες μας αυξήθηκαν με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, γι' αυτό και ε, θεωρούμε ότι πρέπει να μα λάβει υπόψη του και το Κοινοβούλιο φυσικά και τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα. Αποφασίσαμε να καθορίσουμε και τον αναπληρωτή για τους μη εγγεγραμμένους ε, για τη συνεδριάση των συντονισμών. Ε, Όσον αφορά τώρα για τους ε, βοηθούς, αυτοί θα ενημερωθούν απευθείας από τον Ευρωβουλευτή. Καθορίσαμε και ένα σχέδιο χρονοδιαγράμματος για τις ακροάσεις των επιτρόπων και εδώ θα αποστείλω σχετική επιστολή στον ε, πρόεδρο Μπούζεκ διότι σε σχέση με το παρελθόν ε, δεν υπάρχει αποκλειστικός εκπρόσωπος της Επιτροπής ε, Αναφοράς για την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Ο αρμόδιος επίτροπος θα είναι ο επίτροπος σε θέματα οικονομικών η λύση αυτή του να λαμβάνονται υπόψη ε, από κοινού τρει επιτροπέ δεν μα αρέσει, διότι θεωρούμε ότι η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού θα πρέπει να έχει προτεραιότητα στι σχέσει με την Επίτροπο. Καθορίστηκε και ένα χρονοδιάγραμμα για τι επόμενε συνεδριάσει, η οποία ε, θα γίνουν 25 και 26 Ιανουαρίου, αλλά θα πρέπει ίσω να αφήσετε το πρόγραμμά σα ελεύθερο για τι 28 Ιανουαρίου, γιατί μπορεί να πρέπει να κάνουμε μια έκτακτη συνεδρία τη Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού. Τα είπα πολύ γρήγορα, διότι δυστυχώ μα έχει μείνει μόνο μία ώρα στην την οποία πρέπει να συζητήσουμε τρεις ειδικέ εκθέσεις του ελεγκτικού συνεδρίου. Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλώ έχετε λίγο κατά νου τους ε, χρόνους, 20 λεπτά για κάθε έκθεση. Θα ήθελα να ζητήσω και από τους εκπροσώπους λοιπόν του ελεγκτικού συνεδρίου να είναι λίγο πιο γρήγοροι και πιο ακριβείς ε, και λακωνικοί και από εκεί και πέρα θα δούμε αν έχουμε χρόνο για να μιλήσουν και οι συνάδελφοι. Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος. και ελπίζω αυτό να μας εξοικονομήσει και κάποιο χρόνο. Καταρχάς σας ευχαριστώ για τη χθεσινή μικρή δεξίωση που κάναμε. Ήταν και μια ευκαιρία να συζητήσουμε και λίγο πιο ανεπίσημα. και για το θέμα των απαλλογών για τις ε, για τους οργανισμούς, αν θα κάνουμε έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας. Αυτά όλα ε, τα συζήτησαν και οι συντονιστές. Υπάρχουν και διάφοροι παράγοντες που μας επηρεάζουν και καταφέραμε να διευκρινίσουμε και κάποια θέματα. Και συνεπώς, επειδή μίλησε και με τη γραμματεία και ε, μας είπαν ότι υπάρχει και πρόβλημα χρόνος προς τις μεταφράσεις, Ήθελα απλώς να σας ενημερώσω ότι από πλευράς μας άκουσα και κάποιες άλλες πολιτικές ομάδες να έχουν την ίδια άποψη. Συμφωνούμε για τα όσα αποφασίσετε για την έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας για τους οργανισμούς. Ένα ακόμα θέμα στο φάκελό μου έχω και μία πρόσκληση από το Ολλανδικό Κοινοβούλιο για ένα διακοινοβουλευτικό σεμινάριο για τα θέματα του ελέγχου του προπολογισμού. πάντα στο γενικότερο προέσιο των αλλαγών που θα προκύψουν από τη συνθήκη της Λισαβόνας ε, για τη συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Επομένως νομίζω ότι θα ήταν ενδιαφέρον και εδώ λέγεται ότι για κάθε κοινοβούλιο μπορούν να ε, συμμετάσχουν τέσσερις ε, εκπρόσωποι. Επομένως αφορά και εμάς. Φαντάζομαι ότι και εσείς θα λάβατε τη σχετική πρόσκληση. Θα μπορούσαμε ίσως να το συζητήσουμε και να δούμε τη σύνθεση της ομάδας της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου. Ωραία να το αναθέσουμε στη γραμματεία να μας πει δύο-τρία πράγματα παραπάνω και μετά θα το αποφασίσουμε και στις άτυπες συναντήσεις μας. Ευχαριστώ τον κύριο Γκέγερ Να δώσω τώρα το λόγο στο σημείο 9 της ημερήσιας διάταξης ε, στον εκπρόσωπο του ελεγκτικού συνεδρίου, το Μάσιμο Βάρη, τον οποίο θα μας μιλήσει για την ειδική έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου αριθμός 8 κάθετος 2009, δίκτυα αριστείας και ολοκληρωμένα έργα της κοινοτική πολιτικής έρευνας. Επιτεύθηκαν οι στόχοι. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση που σας παρουσιάζει σήμερα το ελεγκτικό συνέδριο έχει αντικείμενο δύο εργαλεία, τα δίκτυα αριστείας και τα ολοκληρωμένα προγράμματα και τα δύο προβλέπονται στο έκτο πρόγραμμα πλαίσιο που χρηματοδότησε την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη 2002-2006 με κονδύλια άνω των 17 δις ευρώ. Αυτή η έκθεση εντάσσεται σε μια συνεχή γραμμή δράσης όσον αφορά προηγούμενα έγγραφα του ελεγκτικού. Παίρνουμε χάρη το 1-2004 για το 5ο πρόγραμμα πλαίσιο και το 9 του 2007 για την εξολόγηση των, της έρευνας που χρηματοδοτείται με κοινωτικά κονδύλια. Τα βασικά προβλήματα στα οποία προσπάθησε να δώσει απάντηση το ελεγκτικό είναι τα εξής. Η Ευρώπη τόνωσε επενδύσεις επαρκώς σε σχέση με την πρόκληση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και οι επενδύσεις που έγιναν διόρθωσαν τις διορθωτικές ατέλειες της ευρωπαϊκής έρευνας. Όπως ξέρουμε, αυτά καλύπτονται και τα δύο από το έκτο πρόγραμμα πλαίσιο. Από τη μια πλευρά το πρόγραμμα προσπαθεί να τονώσει τις επενδύσεις προκειμένου να υλοποιηθεί η μερίστη διάταξη της Λισαβόνας με στόχο τη έρευνα 3% του ΑΕΠ το 2010. Ο ιδιωτικό τομέα τα δύο τρίτα των νέων επενδύσεων. Το πρόγραμμα επίσης θέλει να πετύχει ένα ευρωπαϊκό χώρο έρευνας, ένα σύστημα. Μέσω αυτών των δύο νέων εργαλείων που ανάφερα πριν, δίκτυα αριστείας και ολοκληρωμένα προγράμματα. Τα δίκτυα αριστείας συχνά συνδέουν, συνδυάζουν τους καλύτερους πόρους και εξπερτής σε ένα συγκεκριμένο χώρο για να έχουμε κοινά προγράμματα έρευνας με στόχο μια ενοποίηση των ικανοτήτων των ερευνητών. Έπειτα έχουμε τεχνικές, τεχνικούς, οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους όλοι μαζί προκειμένου να πετύχουμε καινοτομίες σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Γιατί το ελληνικό συνέδριο επέλεξε αυτά τα δύο εργαλεία. Πρώτον, διότι τα σχετικά προγράμματα πιο άμεσα μπορούσαν να βοηθήσουν να δημιουργηθεί αυτός ο ευρωπαϊκός χώρος έρευνας. Δεύτερον, διότι περίπου αποτελούν το 50% του έκτου προγράμματος. Τρίτο, διότι τέτοια εργαλεία μπορεί να χρηματοδοτήσουν πάρα πολλές διαφορετικές ερευνητικές δραστηριότητες από την βασική έρευνα μέχρι την εφαρμοσμένη στους 7 θεματικούς τομείς που έχουν προτεραιότητα. Τι χρηματοδοτήσαμε. Το έκτο πρόγραμμα πλαίσιο χρηματοδότησε 167 προγράμματα δικτύων αριστείας για 5.000 άτομα κοινωτική συμβολή 1,2 δις σε σχέση με 1,9 δις συνολικών επενδύσεων. Κατά μέσο όρο κάθε δίκτυο έχει 30 εταίρους και 7 εκατομμύρια ευρώ εκ μέρους της Ένωσης. Μέσω του εργαλείου των ολοκληρωμένων προγραμμάτων χρηματοδοτήθηκαν 700 πρωτοβουλίες, 17.000 συμμετέχοντες, κοινοτική συνεισφορά 6,5 δις. Μέσος όρος κατά πρόγραμμα 25 εταίροι 9,5 εκατομμύρια ευρώ. Τι λέει η έκθεσή μας. Έχει και θετικά και αρνητικά σημεία. Δηλαδή από μια μεριά να γνωρίζουμε ότι αυτά τα δύο εργαλεία συνέβαλαν στο γενικό στόχο συνεργασία μεταξύ των ερευνητών με αξιόλογα επιστημονικά αποτελέσματα και μια έρευνα για ικανοποίηση που έκανε το ελεγκτικό συνέδριο το επιβεβαιώνει αλλά όταν πάμε να δούμε αν πετύχαμε τους συγκεκριμένους στόχους οι διαπιστώσεις είναι λιγότερο θετικές δίκτυα αριστείας. Γενικά είχαμε συντονισμό των δραστηριοτήτων, είχαμε νέες γνώσεις, μετεφέθησαν οι γνώσεις, οι καινούργιες και οι παλιές προς τη βιομηχανία και προς τους συμμετέχοντες, αλλά οι περισσότεροι εταίροι διέθεσαν στο δίκτυο ένα μικρό ποσοστό των ερευνητικών εκατοντήτων τους και δεν δέχτηκαν η δομή governance του δικτύου να έχουν προτεραιότητα όσον αφορά την χρήση των κοινών πόρων. Μόνο μια μειοψηφία των δικτύων πιστικά κινήθηκε προς μια ικανοποιητική και αυτάρκη ενοποίηση όσον αφορά τους κοινούς πόρους που να έχει δηλαδή προοπτική επιβίωσης μακροπρόθεσμα χωρίς να εξαρτάται από περαιτέρω κοινωτικέ ενισχύσεις. Τα ολοκληρωμένα προγράμματα πετύχαμε την κρίσιμη μάζα για να έχουμε τις καινοτομίε που θέλαμε, ωστόσο αυτό που περιμέναμε την δράση μοχλός στις ε, μέσω των χρηματοδοτήσεων δεν επετεύχθη ούτε ο ρόλος του καταλήτη για το ιδιωτικό κεφάλαιο, ούτε μεγαλύτερη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και σας θυμίζω ότι το έκτο πρόγραμμα πλαίσιο απριόρι έδινε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις το 15% τουλάχιστον του προπολογισμού για τις 7 θεματικές μονάδες. Και τη στιγμή που μειώνεται η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, όπως βλέπετε στους πίνακες που είναι συνημένοι στο κείμενό μας, οι μικροσές επιχειρήσεις δεν ξεπέρασαν καν στη συμμετοχή το 10% και για αντικειμενικούς λόγους και δυσκολίες, αλλά και διότι αποτρεπτικά υπήρξαν εμπόδια στην είσοδο, πολυπλοκότητα, κόστος διαδικασίας να υποβληθούν οι αιτήσει χρηματοδότησης, διάφοροι δεσμοί συμβατικής δομής μακράς διάρκειας, η αυτόματη πρόσβαση στις προηγουμένως γνωστές γνώσεις που το είχαν οι άλλοι εταίροι και η συνολική κοινωνική ευθύνη έναντι της Κομισιόν. Με δύο λόγια, η πρόοδος προς το στόχο να τονωθούν οι επενδύσεις για την έρευνα, τα αποτελέσματα δηλαδή είναι μέτρια. Και η ίδια η Κομισιόν το αναγνωρίζει στα κείμενά της. Η Ευρώπη παραμένει κάτω από το 2% του ΑΕΠ. Βέβαια αυξήθηκαν τα κονδύλια, αλλά η οικονομική συμμετοχή των εταίρων, δηλαδή οι ίδιοι πόροι, για κάθε πρόγραμμα παραμένουν χαμηλοί. Σε μερικέ περιπτώσει υπάρχει αμφιβολία. Η κοινοτική χρηματοδότηση μήπω τυχόν υποκατέστησε τους ιδιωτικούς πόρους, ιδιαίτερα τους δημόσιους. Ο δείκτης από την έκθεση, από τη, στη σχέση συνολικέ επενδύσεις κοινοτική συμβολή μειώθηκε στο έκτο πρόγραμμα σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα πλαίσιο. Το ηλεκτρικό συνέδριο διερωτάται η διαχείριση της Κομισιόν επηρέασε την μερική αυτή επιτυχία των νέων εργαλείων. Στην αρχική φάση ιδιαίτερα το ελεγκτικό επεσήμανε ότι δεν υπάρχει επαρκή σαφήνεια σχετικά με τον ειδικό ρόλο και τη λειτουργία του κάθε εργαλείου σε σχέση με τους στόχους. Πολλές φορές τον, λόγο, ρόλο αυτό δεν τον καταλαβαίνουν όλοι οι εταίροι. Οι συντονιστές λίγο καλύτερα από τους άλλους. Έπειτα η διαδικασία διαπραγμάτευσης πριν καταλήξουμε σε μια υπογραφή συμβολέου κατά τη γνώμη του ελεγκτικού ήταν μακρά περίοδος. 13 μήνες κατά μέσο όρο και έχει πάντα διαφανείς επιπλέον δεν υπάρχει μια λογική παρέμβαση σαφής και ορισμός των στόχων που δυσκόλεψαν την εποπτεία της απόδεσης και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Πορίσματα και συστάσεις εκ μέρους του ελεγκτικού συνεδρίου. Μία σύσταση που την κάναμε και στο παρελθόν τα προγράμματα δαπάνης θα πρέπει να στηρίζονται σε μια συγκεκριμένη λογική, να συνδέει τα εργαλεία με επιτεύξιμους στόχους. Η Κομισιόν για τα δίκτυα αριστείας θα πρέπει να δει προγράμματα συνεργασίας που το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο υποκατέστησε με ολοκληρωμένα προγράμματα και επαναλαμβάνω με ρεαλιστικούς στόχους και με σημαντικά αποτελέσματα σε σχέση με κλασική συνεργασία και αντίστοιχα εργαλεία στην έρευνα. Δεύτερο, η Κομισιόν θα πρέπει να δει τους διάφορους λόγους, ειδικά για το πρόγραμμα πλαίσιο και όχι, που δημιουργούν και χαμηλό επίπεδο επενδύσεων, αλλά και τότε δεν επιτεύχθη η δράση καταλήτη για τον ιδιωτικό τομέα και πιο συγκεκριμένα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τρίτο και τελευταίο, η Κομισιόν πρέπει να βελτιώσει τη διαχείριση των προγραμμάτων, εγγυόμενη σαφής και έγκυρους προσανατολισμούς, πιο γρήγορες διαδικασίες για τις επενδύσεις και καλύτερη υποπτία των προγραμμάτων προκειμένου να αξιολογηθεί η ποιότητα και η επίπτωση των αποτελεσμάτων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η κυρία Γκρέσλη, συγγήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Εκτενέστατη παρουσίαση και θα είμαι σύντομη εγώ γι' αυτό. Και να στήσω σε όλους σας να κοιτάτε τις συστάσεις μας. Προσπάθησα να δω ποιες είναι οι εμπειρίες μας στο παρελθόν και ποιες είναι οι επικρίσεις για την πρόθεση της έρευνας και να τα συνδυάσω όλα αυτά. Είναι πολύ καλή έκθεση πραγματικά και ευχαριστώ το ελεκτικό συνέδριο και την ενημερωτική συνομιλία που είχαμε. Ήταν πάρα πολύ καλή συνεργασία με τον κύριο Βάρη και τους συνεργάτες του άψογη και καλούμαστε το γεγονός ότι αυξάνεται ο προϋπολογισμός της έρευνα να είμαστε και πάρα πολύ προσεκτικοί με σύνεση να κοιτάμε το θέμα. Γιατί τα προβλήματα συσσωρεύονται τα τελευταία 10-15 χρόνια και οξύνονται. Και αν συνεχίσουμε σίγουρα δεν πρόκειται να φτάσουμε στα επιθυμητά αποτελέσματα και αυτά που μας χρειάζονται. Και προσπάθησα να ενώσω όλες τις πηγές, ας πούμε, και την εμπειρία και άλλες πηγές για να ε, δώσουμε τις ε, αιτήσει και τι επιθυμίε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα ήθελα να μα απαντήσει. Πρέπει να σα πω ότι στο έγγραφο εργασία θα κάνω μερικέ μικρέ όμω αλλαγέ που τώρα μόλι ε, υπέπεσαν στην αντίληψή μα. Ε, κάποια γλωσσικά, κάποιε λεπτομέρειε και κάποιε αποφάσει χτεσινέ τη Επιτροπή Ελέγχου για τη διαδικασία ανάκτησης και πριν φτάσουμε στην Ολομέλεια θα ε, χτενίσουμε ξανά το κείμενο. Αυτά τα όλοι είχα να σας πω και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία. Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Γκρέσλε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι είναι. Υπάρχει λοιπόν εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλώ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Ξέρω ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο, γι' αυτό θα εστιάσω σε ελάχιστα σημεία. Ευχαριστώ τον εκπρόσωπο του Ελεκτικού Συνεδρίου και του συναδέλφου του για την πολύ καλή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την κυρία Γκρέσλε για τι πολύ καρποφόρε συζητήσει που κάναμε. Επειδή είπαμε ότι δεν έχω χρόνο, θα εστιάσω σε κάποια θέματα που ανέφερε η κυρία Γκρέσλε στην έκθεσή της. Το ένα αφορά τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να επισημάνω εδώ στα μέλη ότι οι προτινόμενες διορθώσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν προκύπτουν από την εφαρμογή νέας ερμηνείας, αλλά από τις ε, δηλώσεις που υποβάλλουν οι ίδιοι οι χρηματοδοτούμενοι και Αυτό είναι βάση και κανόνων, διότι μπορούμε ακόμα να εποπτεύουμε τα προγράμματα πέντε χρόνια μετά την ολοκλήρωσή τους. Κοιτάζουμε τι δεν είναι ασαφές, συμφωνούμε απολύτως με τη δήλωση και του ελεγκτικού συνεδρίου και, του, και της εισηγήτριας και Δυστυχώ η παρακολούθηση ε, είναι μεγάλο γραφειοκρατικό άθος και για μας και για τους επιδοτούμενους. Επομένως, ε, θεωρούμε ότι η απλούστευση στη διαδικασία ανάκτησης των ποσών και όχι μόνον θα πρέπει να ολοκληρωθεί και εξετάζουμε και τη δυνατότητα μετά από τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ε, μειώσουμε τη διαδικασία για την ανάκτηση των ε, οφειλών. Να ευχαριστήσω και την κυρία Γκλέσσερ, ε, διότι ακολούθησε ακριβώς την ίδια φιλοσοφία με μας. Ο εκπρόσωπος του ελεκτικού συνεδρίου αναφέρθηκε σε κάποιες ελλείψεις ε, στα δίκτυα και στην διαδικασία και εμείς μιλήσαμε με τον καθηγητή Όλμπαρτ και έχουμε σχετική έκθεση και υπάρχουν κάποιες συστάσεις και συμπεράσματα τα οποία συνάδουν με τα συμπεράσματα του ελεκτικού συνεδρίου. Να σας πω όμως ότι η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου αναφέρεται μόνο στο 2006 να πω ότι εμείς έχουμε κάνει κάποια πρόοδο έκτοτε, στο έκτο πρόγραμμα πλαίσιο, συγγνώμη, ενώ για το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο έχουμε κάνει κάποιες διορθώσεις και έχουμε γίνει και μία πολύ σύντομη εξωτερική διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους για το τι μέλη γενέστε με αυτά τα δίκτυα αριστείας. Ξέρουμε ότι αυτό... Ε, συζητήθηκε και στα, στις κοινότητες κοινή έρευνα. Δεν έχουμε καταλήξει ακόμα κάπου. Έχουμε συμφωνήσει βέβαια όλοι ότι πρέπει να υπάρχει δέσμευση για την ολοκλήρωση. Αυτή ήταν η μία παρατήρηση και της έκθεσης του καθηγητή. Και επίσης έχω δύο λεπτά να σας πω και κάποια πράγματα για την απλούστευση. Ναι, σας ευχαριστώ λοιπόν. Για την απλούστευση να υπενθυμίσω στην Επιτροπή σας ότι έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε κάποιες βελτιώσεις στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιων. επαναλαμβάνω, δεν έχουν επιληθεί όλα τα θέματα, φυσικά και όχι. ανέφερε και κάποια στοιχεία η κυρία Γκρέσλε από αυτού. Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ε, το Ταμείο Εγγύσεων, το οποίο μας επιτρέπει να μειώσουμε τον αριθμό ε, αρκετών ελέγχων εκ των προτέρων. Στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο ζητήσαμε πολύ λιγότερα πιστοποιητικά στις ε, οικονομικές δηλώσεις, διότι έχουμε ένα κατόφλι το οποίο εισήγαγε ο νομοθέτης για τις... και υπάρχει συγκεκριμένο ποσό. Κατά πάσα πιθανότητα οι περισσότεροι δεν θα χρειάζεται να δίνουν ένα τέτοιο πιστοποιητικό πλέον και έτσι ε, μειώθηκαν τα πιστοποιητικά κατά 10. Παλιά ζητούσαμε 20 πιστοποιητικά και τώρα κατά μέσο όρο ζητούμε 2. Επίσης έχουμε, κάνει, έχουμε μειώσει τους εκ των προτέρων ε, οικονομικούς ελέγχους. Οι περισσότεροι ε, όσοι ζητούν πάνω από 500.000 ευρώ συνεισφορά θα ελεγχθούν Αυτό σημαίνει όμως ότι 9 στους 10 συμμετέχοντες στο 7ο πρόγραμμα προέλευση θα εξαιρούνται αυτών των εκ των προτέρων ελέγχων. Επίσης έχουμε δημιουργήσει την ενία εγγραφή των συμμετεχόντων και υπάρχει και ένα υποστηριστικό μέσο και έτσι δεν χρειάζεται κάθε φορά που συμμετέχουν να δίνουν ε, τα ίδια στοιχεία, θα τα δώσουν μία φορά και αυτά θα ισχύουν για πάντα. Στην αρχή υπήρχαν κάποια προβλήματα στην εγγραφή, ε, έπρεπε να γίνει μια πρώτα ε, έρευνα, αλλά έχει γίνει πλέον για την όλη διάρκεια ε, του προγράμματος. Έχουμε πλέον 15.000 εγγραφές και υπάρχει ένα και μοναδικό σημείο επαφής. Αυτό ε, διευκολύνει τη διαδικασία και τη συμμετοχή και επίσης επιτρέπει την καλύτερη ποιότητα των δεδομένων. Υπάρχει και μια έκθεση διαχείρισης και προς εσάς αλλά γίνεται και για μας. Έχουμε επίσης εξορθολογήσει όσο γίνεται περισσότερο τον τρόπο για την ανάθεση των ε, συμβάσεων. Έχουμε εξορθολογήσει τον, ε, τις εκθέσεις, έχουμε διευκρίνει τη διάρκεια των προγραμμάτων για τις εκθέσεις στους 18 μήνες και έτσι ζητάμε λιγότερα από τους επιδοτούμενους. Στο 7ο πρόγραμμα πλαίσεων έχουμε μειώσει κατά 40 ημέρες το, τον αριθμό των ημερών σε σχέση με το έκτο πρόγραμμα πλαίσιο. Δεν έχουμε φτάσει βέβαια στο τέλειο, αλλά έχουμε κάνει μία βελτίωση. Και επίσης το χρονοδιάγραμμα για ανάλογα προγράμματα όπου έχουμε πολλούς επιδοτούμενους ε, είναι ένας χρόνος για το χρόνο επαφής. Αυτό ισχύει για παράδειγμα για το ε, Ινστιτούτο Υγείας. Ε, δεν ε, έχουμε τελειοποιήσει τα πράγματα, αλλά έχουμε κάνει καλή δουλειά. Θα σταματήσω εδώ. Υπάρχει ένα ακόμα πράγμα, το είπε και η κυρία Γκρέσλε, το ένα, μία μόνο για όλους. Έχουμε φτιάξει λοιπόν ένα πρόγραμμα πλαίσιο βάση ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουμε μία δικτυακή πύλη και όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν να μπουν σε αυτή τη δικτυακή πύλη και να μπουν στο πρόγραμμα πλαίσιο ανεξάρτητα από το σε ποια γενική διεύθυνση θέλουν να απευθυνθούν. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά το ελεγκτικό συνέδριο και την κυρία Γκρέσλε. Θα τα σημειώσουμε όσα μας είπαν και θα προσπαθήσουμε να βελτιωθούμε περαιτέρω. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν κάποιος θέλει να παρέμβει, αλλιώς να περάσουμε στο σημείο 10. Ειδική έκθεση 14-2009 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα εργαλεία για τη διαχείριση της αγοράς του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων. Επετεύθηκαν οι κύριοι στόχοι. Εκπρόσωπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Γιούλιους Μολνάρ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Δεν θα επεκταθώ σε μεγάλες λεπτομέρειες. Έχετε το έγγραφο εργασίας κυρία Σαλτεμόζε. δεν θέλω να το αναλύσω. Μόνο να κάνω κάποιες ευκρινήσεις σε τρία σημεία. Πρώτον, να σας δώσω ε, σύντομα κάποια στοιχεία για τον λογιστικό αυτό έλεγχο, να σας πω στη συνέχεια τις διαπιστώσεις μας και τέλος τι ε, συνιστούμε και τι συστήνουμε. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της έρευνας, Πρέπει να σας πω ότι η αγορά γαλακτός είναι σημαντικό τμήμα ε, της κοινή γεωργικής πολιτικής, οπότε είναι φυσιολογικό να κάνει το ελεκτικό συνέδριο τακτικούς λογιστικούς ελέγχους. Όπερ και αγέννητο το 2001, σε ειδική έκθεση για το σύνολο της διαχείρισης, του συνόλου μάλλον, των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων. Πέρσι, το 2008, ε, βάλαμε ε, ε, μια νέα έκθεση, ειδική έκθεση για τις γαλακτοκομικές προσθώσεις 10 νέες χώρες που μπήκαν στην Ένωση το 2004. Ο κύριος Χατζημαρκάκης ήταν εισηγητής της ειδικής αυτής έκθεσης, της οποίας, στην οποία επιφυλάξετε πολύ ευνοϊκή υποδοχή. Υποστηρίξτε τότε τις προτάσεις του κυρίου Χατζημαρκάκη και σύσταση, τη σύσταση του συνεδρίου και καλέσει στη συνέχεια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεωρήσουν τα ε, μεταβατικά μέτρα και μέτρα συνοδευτικά που πρέπει να ληφθούν στις περιοχές που κυριαρχούν μικρή παραγωγή ε, μικρές εκμεταλλεύσεις και πρέπει επίσης η γαλακτοπαραγωγή να έχουν όπως είπατε και παραθέτω ένα σταθερό πλαίσιο με ε, σαφείς προοπτικές για να μπορούν να κάνουν τις ζωτικές τους επενδύσεις για να είναι βιώσιμη η εκμετάλλευσή του και η δραστηριότητά τους. Ήδη λοιπόν από το 2001 η ίδια ομάδα έκανε την έκθεση αυτή και το λογιστικό έλεγχο, αλλά πλέον ε, στο σύνολο της διευρυμένης Ευρώπης. Τι διαπιστώσαμε τότε. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα με τους στόχους της ε, κοινής γεωργικής πολιτικής στον τομέα του γάλακτος, καταλήξαμε σε κάποιες διαπιστώσεις αλλά επίσης εντοπίσαμε και παράγοντες κινδύνου που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στη διαδικασία της ε, απελευθέρωσης της αγοράς που ακολουθείται αυτόν τον καιρό. Στραμμένοι λοιπόν προς το παρελθόν, διαπιστώσαμε πρώτα ότι τα εργαλεία της διαχείρισης εμέρι μόνο βοήθησαν για να φτάσουμε σε αυτούς τους στόχους. Για παράδειγμα, διαπιστώνουμε ότι οι ποσοστώσεις όντως επέτρεψαν να πλαισιωθεί κάπως και να ε, οργανωθεί η παραγωγή, αλλά ε, ένα επίπεδο πολύ υψηλό για να αποφευθεί η υπερπαραγωγή. Επίσης, είδαμε ότι η πτυτικότητα των τιμών ε, σε μεγάλο βαθμό και μεγάλο διάστημα αποφεύθηκε, αλλά οι τιμές παραγωγής μειώνονται σε πραγματικούς όρου, ενώ οι τιμές καταναλωτή δεν σταμάτησαν ποτέ να αυξάνονται. Το μέσο εισόδημα των γαλακτοπαραγωγών δεν μπόρεσε τα τελευταία δέκα έτη να διατηρηθεί, παρά μόνο εις βάρος ε, ε κάποιων παραγωγών εκμεταλλεύσεων που εξαφανίστηκαν αυξήθηκε η παραγωγή και αυξήθηκαν και ενισχύσεις. Ο ανταγωνισμός δεν είναι καλός για τα βασικά προϊόντα που είναι ε, το βούτυρο ή ε, το γάλα σε σκόνη ε, που οι παγκόσμιες τιμές είναι χαμηλές. Αντίθετα, στην μεγάλη προστιθέμενη αξία τα προϊόντα όπως το τυρί δεν έχουν τόσο μεγάλες διακοιμάσεις. Ε, υπάρχουν λοιπόν κίνδυνοι που βαραίνουν τον κλάδο αυτό στα πλαίσια της απελευθέρωσης και το ελεκτικό συνέδριο εντοπίζει τρεις βασικούς παράγοντες που θα πρέπει μάλλον να ληφθούν υπόψη λόγω του δημοσιονομικού, του οικονομικού και κοινωνικού αντικτύπου. Και οι παράγοντες αυτοί είναι η αστάθεια των αγορών, η πτυτικότητα των τιμών που πολύ γρήγορα μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικά πλεονάσματα η επιτάχυση της αναδιάρθρωσης με κίνδυνο μιας ε, όλος και μεγαλύτερης ε, γεωγραφικής συγκέντρωσης της παραγωγής και εξαφάνιση πολύ μεγάλου αριθμού παραγωγών ε, στις μη ευνοημένες περιοχές της υπαίθρου. Επίσης, ε, το θέμα της ανταγωνιστικότητας του τομέα που θα πρέπει να δούμε αν μπορεί να ε, προσαρμοστεί στην παγκόσμια αγορά και όχι μόνο ως προς τις τιμές αλλά και ως προς την ποιότητα των προϊόντων. Αυτά λοιπόν που διαπιστώσαμε και οι κίνδυνοι μας οδήγησαν να ε, κάνουμε κάποιες συστάσεις που φυσικά απορρέουν από τα φαινόμενα αυτά. Και τα συνοψίζω ως εξής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εποπτεύει την εξέλιξη της αγοράς για να αποφευθεί κυρίως η επανεμφάνιση μαζικών πλεονασμάτων. Η ε, διαμόρφωση των τιμών παραγωγού και καταναλωτή στο γαλακτοκομικό τομέα θα πρέπει να παρακολουθούνται, γιατί όλο και περισσότερο βάρος έχουν οι μεταποιητές και τα δίκτυα διανομής θα πρέπει να υπάρξουν στρατηγικές για να αντιμετωπιστεί ο διπλός κίνδυνος της ε, γεωγραφικής συγκέντρωσης παραγωγής και της εξαφάνισης των παραγωγών σε ορεινές και μειονεκτούσες περιοχές. Ο προσανατολισμός της παραγωγής προς την ικανοποίηση πρώτα της εσωτερικής αγοράς και για την παγκόσμια αγορά να πάμε προς την παραγωγή ε, προϊόντων υψηλής υπεραξίας όπως είναι το τυρί. Αυτά διαπιστώνουμε και αυτά συνιστούμε. Υπό την έννοια αυτή λοιπόν για να αποφευθεί κάθε παρεξήγηση θα πρέπει να πούμε ότι το τμήμα 6 σχόλια και συστάσεις του εγγράφου εργασίας αποδίδει ε, στο συνέδριο ε, απόψεις που δεν ε, έχει εκφράσει ποτέ και δεν συμμερίζεται ούτε τις αναφέρει στην έκθεσή της. Στο σημείο 1 λοιπόν δεν λέει πουθενά στην ειδική της έκθεση ε, το ελεγκτικό συνέδριο ότι υπάρχει ένας και μοναδικός τρόπος για να εγγυηθούμε τη ε, ισορροπία των αγορών, τη σταθερότητα των τιμών κτλ. Στο σημείο 2. Σε καμία περίπτωση δεν είναι πρόθεση του ελεκτικού συνεδρίου να δημιουργήσει σύγχυση. Αντίθετα, εμείς θέλουμε με τρόπο μερόληπτο να ε, ρίξουμε φως στη συζήτηση και στα διακυβεύματα. Στο σημείο 3 εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι οι γαλακτοκομικές ποσοστώσεις και η ενίσχυση στη Γεωργία θα πρέπει να είναι ένα εργαλείο ανάπτυξης των μειονεκτικών περιφερειών. Στο σημείο 4, το νόημα και το μήνυμα για μας είναι ότι η εσωτερική αγορά είναι οι βασικοί ε, αποδέκτες γιατί μέχρι σήμερα οι εξαγωγές μας αφορούσαν ε, κυρίως βιομηχανικά προϊόντα, βασικά προϊόντα που είναι μη ανταγωνιστικά. Βεβαίως εμείς ε, ενθαρρύνουμε το γαλακτοκομικό τομέα να συμμετέχει στην παγκόσμια ε, κούρσα του ανταγωνισμού, αλλά θα πρέπει να είναι υψηλή ποιότητα τα προϊόντα, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει να ορθοποδήσει και να σταθεί στη διεθνή αγορά. Βεβαίω, εναπόκειται στον εισηγητή και ε, στην Επιτροπή σας, στην εισηγήτρια μάλλον, να κάνει τις συστάσεις και τους προσανατολισμούς και να καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει προτάσεις. Το ελεκτικό συνέδριο δεν έχει κανένα λόγο να αναμειγνύεται στη συζήτηση αυτή. Γι' αυτό θα σας ήμουν ευγνώμων, ανεξάρτητα από τη στάση που θα κρατήσετε και τη στάση που θα κάνετε, να ε, ε, αναλαμβάνετε τις ευθύνες σας, αλλά μην αποδίδετε στο ελεκτικό συνέδριο πράγματα που ποτέ δεν είπε Είμαι ε, στη διάθεσή σα με του συνεργάτε μου και ιδιαίτερα τον κύριο Φένεση που είναι ο Διευθυντής της Ομάδας Λογιστικού Ελέγχου. Και ε, στη διάθεσή σα επαναλαμβάνω για να σα απαντήσω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, το σημειώνουμε. Ο εισηγητή Σαλντεμό έχει το λόγο. Η εισηγητριά μα. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω το ελεκτικό συνέδριο. Πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση του και πάρα πολύ χρήσιμη. Για βέβαια έχω κάποια σχόλια. Και από τις συστάσεις μου φαίνεται αυτό. Φυσικά και χαιρόμαστε που πήραμε έκθεση η οποία αναλύει τον κλάδο και είναι για μας ένα πολύτιμο εργαλείο στο Κοινοβούλιο αλλά και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποθέτω. Διότι η γεωργική πολιτική θα πρέπει να ε, συνεχίζει να μεταρρυθμίζεται μέχρι το έτος 2013. Ταυτόχρονα όμως θέλω να σας πω ότι την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου την αντιλαμβάνομαι κατά πρώτο λόγο ως συνεισφορά στη συζήτηση, ως πολιτικό πλαίσιο, ε, ως ένα μπούσουλα να δούμε πώς ε, μπορούμε να αναπτύξουμε στο μέλλον τη γεωργική πολιτική. Δεν διαφωνώ εγώ με το Ελεκτικό συνέδριο. Και βέβαια θα πρέπει η ευρωπαϊκή αγορά να παρακολουθεί την αγορά και την εξέλιξη των τιμών. Δεν είπα τίποτα διαφορετικό. Μα αυτό το κάνει έτσι κι αλλιώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πολύ καλά το κάνει. Πολύ συγκεκριμένα λοιπόν. Ε, δεν ξέρω πώς μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου, αλλά μας υπενθυμίζει ότι υπάρχουν τέσσερις στόχοι για το γαλακτοκομικό τομέα και θα πρέπει να τους ακολουθούμε. Αλλά οι τέσσερις αυτοί στόχοι είναι μέρη αντιφατική. Γιατί θέλουμε, λέει, ισορροπία στην αγορά και σταθερότητα των τιμών από τη μια και από την άλλη λογικό βιωτικό επίπεδο για τους γαλακτοπαραγωγούς. Και ταυτόχρονα να είναι και ε, ανταγωνιστική η γαλακτοπαραγωγή στην Ένωση. Ε, είναι δυνατόν με τρόπο εύκολο να φτάσουμε και στους τέσσερις αυτούς στόχους ταυτόχρονα. Τα λέω αυτά γιατί τώρα προετοιμάζουμε τη μεγάλη μεταρρύθμιση της Γεωργίας για το 2013. Επίσης, εγώ πουθενά δεν λέω ότι λέει ε, κάποια πράγματα το ελεκτικό συνέδριο να καταργηθούν οι γαλακτικές, γαλακτοκομικές ε, συγγνώμη, ποσοστώσεις. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Απλώς λέγω ότι έχουν ήδη ληφθεί πολιτικές αποφάσεις σχετικά. Και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Να μην οδηγηθούμε σε συγχύσεις ανάμεσα στους στόχους της πολιτικής μας ε, ε, για το γάλα και στα υπόλοιπα γιατί οι αγρότες αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες. Θέλω να πω και σε κάποιε λεπτομέρειε τώρα. Σημαντικός ο στόχος, ε, σημαντική η στόγευση, αλλά ακόμα σημαντικότερε οι συνέπειε για τη γεωργία ε, στις ορεινέ περιοχές και στις μειονεκτικέ περιοχές. Τι γίνεται επίση με τι επιδοτήσεις. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να πηγαίνουν οι γεωργικές επιδοτήσεις. Υπάρχουν ε, άλλα κονδύλια που λέγονται ανάπτυξη της υπαίθρου. Και θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε ανταγωνιστικοί στη γαλακτοπαραγωγή. Και δεν θα πρέπει να έχουμε γνώμονα μόνο την εσωτερική αγορά στην Ένωση, όχι, την παγκόσμια αγορά. Και θα πρέπει να είναι και αποδοτικό ο τομέα και κερδοφόρος για να μην σπαταλούμε ε, πόρους των φορολογουμένων. Επαναλαμβάνω, είναι πολύ καλή η έκθεση. Μας θυμίζει τα όσα ε, πρέπει να συζητήσουμε στο μέλλον για τη γεωργία, για τη γεωργική πολιτική και τη μελλοντική τη εξέλιξη. Αλλά θα πρέπει να ανησυχούμε ε, τους αγρότες, να τους προκαλούμε ε, ανασφάλεια. Θα πρέπει να ε, συνεχίσουμε την πολιτική μας, να απελευθερώσουμε το τομέα, αλλά με τρόπο λογικό, καλό, συντεταγμένο και είναι πολύτιμα τα στοιχεία του ελεκτικού συνεδρίου. με βέβαιο ότι ήδη από σήμερα τα εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περιμένω να ακούσω τα ενδιαφέροντα σχόλιά σας πολύ. Λοιπόν, ζήτησαν Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο, διότι κατά την άποψή μου ανέφερε πάρα πολύ σημαντικούς τομείς προβλημάτων που δεν μπορεί να απαντήσει βεβαίω πολιτικά. Ανοίγει τα ερωτηματικά, πραγματικά ε, υπαρκτά και θα ήθελα από την αρχή να παρακαλέσω όλους τους συναδέλφους, ο καθένας έχει τη δική του εμπειρία με τη χώρα του, με τις περιφέρειές του, το περιβάλλον και τη, τους αγρότες του και τους κτηνοτρόφους του και τις οργανώσεις και τις εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να καταλάβουμε ότι στη Γεωργία έχουμε πολύ μεγάλες διαφορές στις περιφέρειες και πολύ μεγάλες διαφορές στις προϋποθέσεις. Για να μπω στα συγκεκριμένα. Αυτή η ανεξέλεγκτη συγκέντρωση πολύ με εντυπωσίασε και πραγματικά είχα την ευκαιρία να το διαπιστώσω αυτό πάρα πολύ καλά. Κυρία Σάλτε Μόζε, κατά την άποψή μου, δεν είναι βέβαιο ότι οι γαλακτοκομικές ποσοστώσεις θα σταματήσουν αυτή την ανεξέλεγκτη ε, συγκέντρωση. Καταστρέφονται ε, μικρομεσαίες ε, επιχειρήσεις κερδοφόρες και αυτό θα μπορούσε να ε, προκαλέσει προβλήματα και δημόσιας υγείας αλλά και προβλήματα περιβάλλοντος και διανομής αν συγκεντρωθούν τα πάντα σε ένα σημείο. Ακριβώς ετίθενται ερωτηματικά που πρέπει να απαντήσουμε και θα πρέπει να συζητήσουμε για τις περιφέρειες αυτές. Εγώ τις γνωρίζω καλά, την, τον Νότιο Ρόλο, την Αυστρία, τη δική μου περιφέρεια, ακόμα και την Ιταλία και παρατηρώ ότι η καταστροφή ακριβώς μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μικρομεσαίων εκμεταλλεύσεων είναι προβληματική γιατί προσανατολίζονται προς την αγορά, την παγκόσμια. Και τελικά δεν βάζουμε, ε, ε, αν δεν καταστρέφαμε αυτές τις επιχειρήσεις δεν θα χρειαζόταν στη συνέχεια να δίνουμε κονδύλια στην ανάπτυξη της υπαίθρου ή στην ανοικοδόμηση των χωριών που ε, ρημώνουν και ρημάζουν ή για τη διάβρωση του εδάφους. Κανένας δεν μπορεί να τα κάνει αυτά καλύτερα από τους ίδιους τους αγρότες. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ενισχύσουμε τις μικρομεσές, τις μεσές ε, εκμεταλλεύσεις, τις αγροτικές ε, και όλα αυτά τα λέει πολύ ωραία η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Στη συνέχεια, πολύ σημαντικό επίσης θεωρώ, αυτό που λέει ε, για την παγκόσμια αγορά η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Χρειάζεται επιγόντως να τα συζητήσουμε και αυτά τα θέματα. Ποια είναι η σκοπιμότητα ε, των κονδυλίων ε, που επιδοτούμε. Θα πρέπει να πουλάμε προϊόντα τα οποία να αντέχουν στο διεθνή ανταγωνισμό και όχι να κάνουμε εξαγωγές για να παίρνουμε τις επιστροφές των εξαγωγών και δεν βοηθάει αυτό κανέναν. Οι κοστίζει πολλά και δεν έχουμε και ανταγωνιστικά προϊόντα. Επίσης θα ήθελα να σας πω και σε σχέση με την ανεξέλεγκτη συγκέντρωση της παραγωγής ότι στο μεταξύ η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας αρχίζει να συζητάει τη μακροπρόθεσμη αποθήκευση τροφίμων γιατί υπάρχει πρόβλημα. Αυτό δεν μπορούν να το κάνουν οι αγρότες γιατί δεν έχουν τις αποθήκες ούτε οι μεγάλες εκμεταλλεύσεις καν. Και αυτό το σκεφτούμε λοιπόν. Συγγνώμη, όχι, προφανώς όχι η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, ο ΦΑΟ. Δεν ξέρω αν τα σημεία 1 και 2 είναι τόσο απαραίτητα στην έκθεση, γιατί ομολογώ ότι και εγώ έτσι τα κατάλαβα, όπως είπε το ελεκτικό συνέδριο. Ούτε δρόμο προτείνει, ούτε σύγχυση προκαλεί το συνέδριο αυτό καθ' αυτό. Το συνέδριο δεν πιστώς έρχεται να κάνει. Τα προβλήματα τα προκαλούν όλα αυτά. Τα προβλήματα της γεωργίας ε, μας έχουν οδηγήσει σε αυτή την αντιπαράθεση, όχι το ελεκτικό συνέδριο. Ευχαριστώ. Grazie. Vi prego eh. Παρακαλώ κρατιέσαι, να κρατιέσαι μέσα στα δύο λεπτά. Housling. Ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ για την έκθεση και την καλωσορίζω και στην Επιτροπή Γεωργίας τη συζητήσαμε ε, συντομία. Βέβαια παραμένουν πολλά θέματα ανοιχτά. Σωστό είναι αυτό. Ας πούμε τι θα γίνει στο μέλλον ε, με την αγορά των γαλακτοκομικών και την καθοδήγησή της και μέσα και τα εργαλεία. Βλέπουμε τι γίνεται αυτό το καιρό όταν έχουμε ανισορροπίες στην αγορά πολύ μεγάλη προσφορά, υπερπροσφορά, πολύ χαμηλή ζήτηση και ο Ευρωπαίος φορολογούμενος έχει ένα σωρό κόστος ε, με την αποθήκευση της επιδοτήσεις ε, στις εξαγωγές και αν το προβάλλουμε αυτό στο 2015 τι βλέπουμε. Ότι δεν είναι απαραίτητο πλεονέκτημα για την ευρωπαϊκή αγορά να μην έχουμε ρυθμίσεις τέτοιες ας πούμε να συνεχιστούν οι ποσοστώσεις. Αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να τα απαντήσουμε κάποια φορά. Και έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σωστά, βέβαια δεν μίλησε ακόμα εδώ, αλλά σωστά μας λέει ότι το ελεκτικό συνέδριο ήδη από το 2001 έχει γνωμοδοτήσει ε, και ε, οδηγεί σε αυτή την απελευθέρωση. Τώρα τι λέει, υπάρχουν νέα στοιχεία ε, που μας οδηγούν να έχουμε ένα πιο επικριτικό πνεύμα και βλέμμα ή πώς έρχεται η νέα αξιολόγηση να απαντήσει την προηγούμενη που λέει ότι στο μέλλον θα εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε μηχανήματα κατεύθυνση καθοδήγηση τη αγορά, να μην την αφήσουμε στη μοίρα τη και πέσει σε ανισορροπίε. Και τι γίνεται με τι μειονεκτικέ περιφέρειε. Όντω, ε, και μέχρι τώρα οι απαντήσει δεν είναι ικανοποιητικέ και δεν μπορούν να χρηματοδοτούνται τα πάντα από το δεύτερο πυλώνα ή να τα διορθώνουμε. Θα χρειάζονται απαντήσει έτσι επί τη ουσία για να λύσουμε τα προβλήματα σε ολόκληρες τις ε, περιφέρειες αυτές. Αυτά. Και βεβαίως δεν πρέπει να είναι αυτός σκοπός η απελευθέρωση. Θα πρέπει να σκεφτούμε τι κάνουμε με διάφορες ε, αγορές ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μήπως χρειάζονται ακόμα ρυθμίσεις. Uh, uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχουμε σήμερα μια πολύ καλή έκθεση, ιδιαίτερα οι συστάσεις. Ε, το γάλα και τα γεωργικά προϊόντα είναι κάτι το αφιλεγόμενο στην Ένωση, ιδιαίτερα δεν προτείνονται αλλαγέ. Το είδα και εγώ ίδιο όταν πήγα διακοπέ στη Γαλλία. Είδα ένα σωρό διαμαρτυρίες για το γάλα. Βέβαια η Ένωση των Αγροτών στο Ηνωμένο Βασίλειο συμφωνεί να πάψουν οι ποσοστώσεις. Δεν έχει πρόβλημα με τον ανταγωνισμό. Επίσης, θα αναγνωρίσουμε ότι η μεγάλη συζήτηση για την γεωργική πολιτική ε, θα γίνει στα πλαίσια του 2013. Ιδιαίτερα η σύσταση που λέει ότι υπάρχει παραπάνω από προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα του γαλακτοκομικού και γεωργικού τομέα, που σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν και άλλε πολιτικές σε σχέση με την Ήπεθρο. Βέβαια, αυτό δεν είναι σημερινό θέμα. Είναι για το μέλλον. Να κάνουμε μια πιο ευρεία συζήτηση για τα θέματα της Ήπεθρο. Τι γίνεται με την φτώχεια στην Ήπεθρο. Ότι η φτώχεια δεν είναι μόνο το εισόδημα, υπάρχουν και άλλες πτυχές είναι η πρόσβαση στις το δίκτυο μεταφορών, η στέγαση και άλλα. Επίσης, όταν μιλάμε για τον προπολογισμό στους επόμενους μήνες, θα πρέπει να δούμε τους διάφορους πυλώνες, άμεσες επιδοτήσεις, ανάψυξη της υπαίθρου, πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση, στη συζήτηση για τον προπολογισμό. Σήμερα κοιτάμε τις συστάσεις και οι στάσεις συμφωνούν, είναι σαφείς. <coughs> Και τώρα στον κύριο Βερστέιλεν της Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. και εμείς επικρατούμε την έκθεση του Ελληνικού Συνεδρίου για να συζητηθούν οι εξελίξεις στο γαλακτοκομικό τομέα. Όπως ξέρετε η πρόκληση για τον τομέα αυτό μας στα πλαίσια της απελευθέρωσης και της παγκοσμιοποίησης είναι να γίνει πιο ανταγωνιστική ή να κλείσει το χάσμα που είχαμε στη διαφορά τιμών 30% με τις διεθνείς τιμές ταυτόχρονα Θέλουμε να κρατήσουμε μια ανταγωνιστική παραγωγή γάλακτος στη, ιδιαίτερα στις πιο ευπαθείς περιοχές της υπέθρωνα. Για να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί, μειώσαμε τις τιμές, μειώσαμε το δίκτυο ασφαλείας και δώσαμε εισοδηματική ενίσχυση 7 δις άμεσες ενισχύσεις με αποσύζευξη αυτή τη στιγμή αλλά έχουν συνδεθεί με την cross compliance. Επίσης προσπαθούμε όσο μπορούμε να βοηθήσουμε τον κλάδο να γίνει πιο ανταγωνιστικός. Επίσης η προσπάθεια είναι να καταργηθούν οι ποσοστό το 2015. Σα θυμίζω ότι το εργαλείο αυτό ξεκίνησε το 1984 ως προσωρινό. Και όλοι συμφωνούμε ότι σε μια απελευθερωμένη αγορά και πιο ενοποιημένη παγκόσμια, το σύστημα των ποσοστώσεων δεν στέκεται. Αυτό λένε και οι συστάσεις του Ελληνικού Συνεδρίου του 2001. Όλοι ξέρουμε ότι ζούμε μια δύσκολη συγκυρία όσον αφορά το γάλα λόγω της γενικότερης οικονομικής κρίσης το 2007 ψηλή ζήτηση, ψηλές τιμές. Αυξήθηκε η ζήτηση και τώρα έχουμε χαμηλές τιμές το 2008. Αυτά μέσα στα πλαίσια μιας σταθερής παραγωγής. Δηλαδή τα δύο χρόνια αυτά είχαμε την ίδια παραγωγή. 4% κάτω από την ποσόσταση, άρα η ποσότητα δεν έπαιξε σημαντικό ρόλο. Ήταν η ζήτηση που μέτρησε, που μειώθηκε και έχουμε το δίκτυο ασφαλείας της παρέμβασης. Το ανοίξαμε και λειτουργήσε. Γιατί αγοράσαμε βούτυρο από βουτυρωμένο γάλα σε σκόνη και ε, επαναφέραμε και το εργαλείο των εξαγωγικών επιδοτήσεων. Οι τιμές σταθεροποιήθηκαν σε επίπεδο δικτύου ασφαλείας και σιγά σιγά άρχισαν να αυξάνονται. με αγορά περίπου το 2% του ισοδύναμου γάλακτος, δηλαδή το ποσά μικρά. Αυτή τη στιγμή, λόγω αυτών των εξελίσσεων και των, περιφερει... ε, ε εποχιακών διακυμάνσεων, οι τιμές για το βούτυρο και το απογοητευμένο γάλα είναι γύρω στο 25% πάνω από την τιμή παρέμβασης. Και αυτό αντικατοπτρίζεται και στις τιμές γάλακτος για τον παραγωγό. Βέβαια, οι τιμές ακόμη είναι 20% κάτω από το ψηλότερο επίπεδο τους πέρυσι. Ζούμε λοιπόν αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Έχουμε την έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου. Και είναι η ερώτηση. Η πολιτική αυτή πρέπει να συνεχιστεί. Μήπως θα έπρεπε να συγκεντρωθούμε περισσότερο στα θέματα εσωτερικής αγοράς και όχι εξωτερικής. Ή επισημαίνει τα μειονεκτήματα της κατάργησης των ποσοστώσεων η έκθεση. Και γίνεται και η σύσταση η Κομισιόν να παρακολουθεί η απελευθέρωση να μην οδηγήσει σε υπερπαραγωγή. Ένα είδος θεσμικής υποπτίας των ποσοτήτων. Ξαναγυρίζουμε στους ποσοστώσεις δηλαδή. Αυτό πρέπει να δημιουργήσει σύγχυση. Γι' αυτό λέμε, ναι μεν καλή η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου, αλλά η έκθεση της κυρίας Σέλντεμος είναι ακόμα καλύτερη, διότι ζητάει από την Κομισιόν να εξακολουθήσει να εφαρμόζει τις πολιτικές αποφάσεις για να μην έχουμε σύγχυση. Επίσης διαβεβαιώνω και την Επιτροπή σας και το Ελληνικό Συνέδριο ότι η Κομισιόν θα κάνει ό,τι μπορεί προδραστικά οι αποφάσεις αυτές να συνοδεύονται με μέτρα αγοράς με την αναδιάρθρωση του πακέτου ανάκαμψης και έχουμε και ομάδα υψηλού επίπεδου που θα συζητήσει τα θέματα αυτά, ιδιαίτερα πώς θα καταπολεμηθεί η άκρα μεταβλητότητα. Στην παραγωγή της αλυσίδα, ιδιαίτερα μεταξύ παραγωγών και μεταποιητών, η διαπραγματευτική εξουσία και δύναμη μάλλον που έχουν οι μικροί παραγωγοί, περισσότερη διαφάνεια, καινοτομίε, ποιότητα, σήμανση και το μέλλον των μέτρων της αγοράς και άλλα εργαλεία όπως futures τα οποία μπορούν να καλύπτουν τον κίνδυνο των τιμών. Η ομάδα που ανάφερα έχει συνδυάσει κάποιες φορές, θα ξανασυνδυάσει το Δεκέμβριο, πάλι τον Ιανουάριο, κάθε τρεις εβδομάδες. Και την έκθεσή μας μάλλον θα είναι έτοιμη τον Ιούνιο του 2010. 26 Μαρτίου θα κάνουμε και μια διάσκεψη όπου όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν μέρος. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε και περνάμε στο σημείο 11. Ειδική έκθεση 10-2009. Ενημέρωση και πρόθεση για τα γεωργικά προϊόντα. Το μέρος του Ελληνικού συνεδρίου Γιώργης να έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πριν σας παρουσιάσω πάρα πολύ σύντομα την έκθεση αυτή, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τον κύριο Φιέλνερ για το έγγραφο εργασία του, το οποίο με τρόπο σαφέστατο ε, σκιαγραφεί την ειδική έκθεση και τα συμπεράσματά του βασίζονται σε μία απόλυτη και πλήρη κατανόηση και γνώση της έκθεσής μας και των συμπερασμάτων. Οπότε δεν θέλω εγώ να αναλύσω τα όσα λέει ο κ. Πιέλνες στο έγγραφο εργασία του. Θα περιοριστώ μόνο στα βασικά σημεία της έκθεσης. Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση υλοποιεί και χρηματοδοτεί δράσεις πρόθεσης γεωργικών προϊόντων ήδη από την αρχή ε, της δεκαετίας του 80. Και αυτό μπορεί να είναι δράσεις δημοσίων σχέσεων, διαφήμιση, προώθηση προϊόντων ε, για να καταδειξεί τα πλεονεκτήματα των κοινοτικών προϊόντων, ας πούμε, ως προς την ποιότητα, την υγιεινή, την επιστημιστική ασφάλεια, την ασφάλεια τροφίμων, τον σεβασμό του περιβάλλοντος. Αυτές λοιπόν οι δράσεις προώθησης ε, είναι στο λεγόμενο πράσινο κουτί των διαπραγματεύσεων του ε, ΠΟΕ και χωράει και περισσότερη ανάπτυξη. Αυτό το καιρό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβληματίζεται σε βάθος για το καθεστώς αυτό που θα ε, μπορούσε να ε, βοηθήσει για να ε, αυξηθεί πολύ ο προπολογισμό για την προώθηση των προϊόντων και τη διαφήμιση. Υπό το πρίσμα λοιπόν αυτό, το ελεκτικό συνέδριο ήλεγξε την αποτελεσματικότητα των δράσεων και την κανονικότητα των δαπανών. Ο έλεγχος αυτός, ο λογιστικός έγινε στις υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στις σε τρεις μεγάλες ε, χώρες μάλλον που είναι βασικοί δικαιούχοι των μέτρων. Και έχουμε καταλήξει σε τέσσερις βασικές διαπιστώσεις και συστάσεις από αυτόν. Τις εξής. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα τελευταία χρόνια άρχισε να βελτιώνει τη διαχείριση και τον έλεγχο αυτών των ε, δαπανών για τα προϊόντα. Αυτή η διαδικασία ε, βοήθησε να έχουμε θετικά αποτελέσματα σε κάποιους τομείς και θα πρέπει και πάλι να επιβεβαιωθεί και να ευαθυνθεί. Στη συνέχεια, το ισχύον σύστημα δεν επιτρέπει να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα της πολιτικής αυτής. Ε, ο αντίκτυπός της, ακόμα και αν είναι θετικός μάλλον, δύσκολο να μετρηθεί. Είναι μεγάλη η φιλοδοξία και για να μετρήσουμε τον προπολογισμό σε σχέση με τη φιλοδοξία θα πρέπει να βάλουμε στόχους και δείκτες ε, επιδόσεων. Ε, μια διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερμένους φορείς θα πρέπει να γίνει έτσι ώστε να υπάρξει μια συνολική στρατηγική και συμπληρωματικότητα με τις διάφορες ε, ισχύουσες και υπάρχουσες δράσεις πρόθεσης. Τρίτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έγινε πλέον πιο επιλεκτική στην έγκριση των ε, προσχρηματοδότηση προγραμμάτων. Τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να συνεχιστούν, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ενημέρωση για ε, τον αντίκτυπο που περιμένουμε από το πρόγραμμα και πώς αυτό θα μετρηθεί. Επίσης, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν να είναι ε, πιο επιλεκτικά. Και τέλος, σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των προγραμμάτων και την κανονικότητα των δαπανών, θα πρέπει να γίνουν πρώτα απ' όλα προσπάθειες για τους ελέγχους που είναι πολύ περιορισμένου ακόμα, τους οργανισμούς εκτέλεσης που παίζουν ρόλο κλειδί. Η μεταγενέστερη και η εσωτερική παρακολούθηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής βελτιώθηκε. Αλλά υπάρχουν σημαντικές αδυναμίες ελέγχου, οι οποίες ε, παραμένουν στα διάφορα κράτη-μέλη και εδώ θα πρέπει να γίνει παρακολούθηση για να έχουμε ε, ταχύτερη διόρθεση των αδυναμιών. Αυτά είναι λοιπόν τα μηνύματά μας. Η άλλη μια φορά, δεν αποκλείεται ο προγραμματισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ε, οδηγήσει σε πρόταση γενναίας αύξησης ε, του προϋπολογισμού διαφήμισης και προώθησης. Εκεί η βελτίωση της ε, διαχείρισης έχει κάθε λόγο ύπαρξη. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος των εισηγητή, ο κύριος Φιέλνερ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καταπληκτικά. Από ό,τι κατάλαβα πρέπει να είμαι σύντομος, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Θα μπορούσα να ξεκινήσω λέγοντας ότι όταν ανέλαβα αυτή την έκθεση, είχα μια προσωπική ιδέα για το πώς λειτουργεί το σύστημα, πολύ πολιτική ιδέα και θα πρέπει να πω ότι είμαι ένας από αυτούς που θα ήθελε να αμφισβητήσει την καταλληλότητα όλη αυτή τη ιδέα του να παίρνουμε τα χρήματα των φορολογουμένων και κατόπιν να τα χρησιμοποιούμε για, να... τα διαφημί... για διαφήμιση για να προσπαθήσουμε να του ξαναπουλήσουμε προϊόντα. Παραδείγματο χάρη, στη Σουηδία ε, διαφημίσεις για ισπανικά πορτοκάλια, ολλανδικούς χυμού ε, και όλα αυτά φυσικά δημιουργούν και διαφιλονικίε και πυροδοτούν και τον ε, σκεπτικισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι βέβαια αυτό το θέμα της συζήτηση, του κατά πόσο είναι σωστό ή λάθος. Ε, ε, κοιτάμε κατά πόσο έτυχαν το στόχο τους και τι γραφειοκρατία υπήρχε στην πορεία. Νομίζω ότι θα πρέπει να συζητήσουμε λίγο την πολιτική για να δούμε κατά πόσον είναι κατάλληλο ή όχι αυτό που κάνουμε. Είναι πολύ σημαντικό διότι είναι πολλά τα λεφτά έχουν διπλασιαστεί, υπερδιπλασιάστηκαν τα τελευταία χρόνια. Έχουμε μία σειρά από προγράμματα τα οποία ε, αυξήθηκαν επίσης στον αριθμό και αυτά διπλασιάστηκαν και ε, μας μιλάτε για βελτιωμένους ελέγχους και καλύτερη διοίκηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ως συνήθως, όπως λέω, πολλά πράγματα ε, περιμένουμε και από την παρακολούθηση των κρατών μελών. Με ικανοποιεί ιδιαίτερα το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, επειδή διαπίστωσε ότι υπήρχαν προβλήματα στην Ισπανία και στην Ιταλία στο παρελθόν, κατάφερε πλέον να ε, συγκρατήσει την κατάσταση και ελπίζω αυτή η τάση να συνεχιστεί στο μέλλον. Αν θέλουμε να προσπαθήσουμε να έχουμε μια εικόνα του κατά πόσον επιτυγχάνονται οι στόχοι σε αυτό το τομέα της πολιτικής, νομίζω ότι είναι προφανέ ότι η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου θα πρέπει να διευκρινίζει ποιοι είναι αυτοί οι στόχοι. Είναι δύσκολο να έχουμε κάποια ορόσημα και, και τι, ε, να ξέρουμε τι μετράμε, αν δεν ξέρουμε με τι πρέπει να τα συγκρίνουμε. Επίση, θα πρέπει να ε, ξέρουμε ότι το επίπεδο φιλοδοξία <coughs> και το επίπεδο των στόχων ε, σχετίζονται το ένα με το άλλο. Όπως λέει η μαμά μου πολύ συχνά, ε, ή κέρδισε τα όλα ή χάσε τα όλα. Αν προσπαθείς να λείψεις ένα τόσο ευρύ φάσμα πραγμάτων, τείνεις να χάνεις τελικά όλο σου το στόχο και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαβάσει και αυτή τα μαθήματά της λίγο. Πρέπει να είμαστε σίγουροι αν είναι κατάλληλος ο προπολογισμό για το επίπεδο φιλοδοξία που προσπαθούμε να επιτύχουμε. Επίσης υπάρχει και το θέμα του κριτηρίου SMART. Ναι, και αυτό είναι κάτι το επισημένο. Θα πρέπει να υπάρχουν κριτήρια τα οποία θα μπορούν να είναι μετρήσιμα και θα μπορούμε να τα παρακολουθούμε. Αν δείτε το θέμα, διαπιστώνετε ότι υπάρχουν κάποιε χώρε που χρησιμοποιούν ε, πάρα πολύ. Προσπαθώ λίγο να το σκεφτώ και με απλά αριθμητικά στο, ε, απλή αριθμητική στο κεφάλι μου. Η Ιταλία και η Ισπανία και νομίζω ε, λίγε άλλε χώρε, ουσιαστικά παίρνουν το 75% όλου αυτού του προγράμματος. Και η ερώτηση μου είναι γιατί. Θα πρέπει να υπάρχει ανταγωνιστικότητα και τα πάνε καλά για την ανταγωνιστικότητα, λαμβάνοντας υπόψη και τα προϊόντα που εγώ ως πολίτης στη Σουηδία μπορώ να έχω γιατί λαμβάνονται λοιπόν αυτά τα μέτρα μόνο σε λίγες χώρες. Θέλω λίγο να το καταλάβω. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ένα λεπτό στο, στην κυρία Σαλτεμόζα και μετά θα ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ. Ναι, θα είμαι σύντομη. Θέλω να πω μόνο ότι υποστηρίζω τον εισηγητή και συμφωνώ με τις παρατηρήσεις του για την έκθεση αυτή. Αλλά υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα ότι δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα αν λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα. Γιατί δεν μπορούμε να μετρήσουμε και τη λειτουργία και τις επιπτώσεις. Αφήστε που διαπλασιάστηκε τώρα το ποσό. Πάντως υποστηρίζω αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ. Για να ολοκληρώσουμε, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, ο κύριος Σωτάτη, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω το ελεκτικό συνέδριο για την αρκετά θετική έκθεση σχετικά με την πολιτική ενημέρωση και προώθηση, καθώς επίσης και τον εισηγητή τον κύριο Φιέλνερ. Θα μπορούσα εγώ να είμαι συντομότατος, διότι το σύνολο των συστάσεων του Ελεκτικού συνεδρίου και του συγητή έχουν σχεδόν αρχίσει να εφαρμόζονται στη νέα πολιτική πρόθεση. Είναι γεγονός ότι διπλασιάστηκε ο προϋπολογισμός, αλλά πρόκειται για αύξηση από τα 23 εκατομμύρια στα 50 εκατομμύρια. Δηλαδή είναι αρκετά λογικό ακόμα το πλαίσιο από την έκδοση της έκθεσης του ελεγκτικού συνεδρίου και ε, το έγγραφο του εισηγητού και μετά τι κάναμε. Είμαστε ακόμα πιο αυστηροί ακριβώς στην επιλογή των προγραμμάτων και θέτουμε το βάρος εκεί που προτείνει και ο εισηγητής και το ελεγκτικό συνέδριο. Δηλαδή, ε, έρευνες αγοράς και αντικτύπου εκ των προτέρων, σαφείς στόχους, ευφυείς, smart, ε, στόχους που να συνδέονται με τις δράσεις και αποτελεσματικές δράσεις και πιο σημαντικό μέθοδο αξιολόγησης που να μας επιτρέπει ετησίως να μετρούμε τον αντίκτυπο και τα αποτελέσματα των δράσεων πρόθεσης. Αν δεν έχουμε τέτοιες δράσεις ε, και τέτοια αξιολόγηση, το πρόγραμμα απορρίπτεται. Ξέρετε ότι στην Ευρώπη έχω τη φήμη εκείνου που απορρίπτω όλα τα προγράμματα διαφήμισης και προώθησης. Απορρίπτονται πάνω από 60% των προγραμμάτων γιατί δεν έχουν εκείνα τα βασικά στοιχεία που να μας επιτρέπουν τη δαπάνη κάθε ευρώ αυτής της πολιτικής ε, προώθησης. Για τη μελλοντική στρατηγική η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προβληματίζεται. Ακόμα δεν έχουμε νέα διότι αλλάζουν καθημερινά ε, οι καταστάσεις και όπως λέει το ελεκτικό συνέδριο δεν είναι βέβαιο ότι θα αυξήσουμε τον προϋπολογισμό για την πρόθεση και την ενημέρωση. Υπάρχουν διάφορες φόρμουλες που συζητούμε και δεν ε, καταλήγουν όλες αυτόματα σε αύξηση ε, του προπολογισμού για την πολιτική πρόθεση προϊόντων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου το απόγευμα. Σας ευχαριστώ πολύ.